Λοιπόν, καλώς ορίσατε, αγαπητοί συνάδελφοι, για την τρίτη ακρόαση που έχουμε σε αυτές τις δύο μέρες. Πρόκειται για τη χρηματοδότηση των πνευματολογικών αλλαγών. Θα πρέπει να οργανωθούμε σωστά για να τελειώσουμε πραγματικά στις 5 μετά τι εμπειρίες των πρώτων δύο ακροάσεων, θα σας να ευγνώμων αν όλοι τηρούσαν το χρόνο που τους έχει χορηγηθεί, για να μπορέσουν έτσι και πολλοί συνάδελφοι να υποβάλουν ερωτήσει και να ακούσουν και απαντήσει. Αυτά εισαγωγικά. Η συνάδελφο Ποδηματά θα ήθελε κάτι να πει εισαγωγικά, νομίζω. Σειρά σα είναι, κυρία Ποδηματά. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρόιλ. Αγαπητοί προσκεκλημένοι κύριε και κύριοι συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην πρώτη αυτή ακρόαση για τη χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής. Οφείλω να ομολογήσω ότι μου ήρθε η ιδέα αυτή της ακρόασης πριν από λίγους μήνες όταν αντικατέστησα τον πρόεδρό μας τον κύριο Ρόιλ σε μια διακοινοβουλευτική διάσκεψη που είχε οργανώσει η Σουηδική Βουλή στη Στοκχόλμη όπου συνάντησα την εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, την κυρία Γκλέιτ, και εντυπωσιάστηκα από αυτά τα οποία μας είπε και τα στοιχεία που μας έδωσε. Βεβαίως τότε υπήρχαν προσδοκίες για μια παγκόσμια δεσμευτική συμφωνία στην Κοπενχάγη και δεν είμαι σίγουρη πως αυτό ισχύει πλέον. Οπότε υπήρχαν κάποια, κάποιες επιφυλάξεις ε, για την οργάνωση μιας τέτοιας ακρόασης ε, δύο εβδομάδες πριν από την Κοπενχάγη που υπετίθετο ότι θα είχαμε καταλήξει σε μια κοινή θέση στα βασικά στοιχεία μια συμφωνίας. Θα ήταν λοιπόν άκερη η διοργάνωση της ακροασίας και μακάρι να ήταν σωστό αυτό, αλλά δυστυχώς 30 μέρες, λιγότερο από 30 μέρες πριν από την επίσημη ένταξη Κοπεχάγης, η συζήτηση που γίνεται στο ευρωπαϊκό και το διεθνές επίπεδο τονίζει πως η απόφαση για την οικονομική πτυχή της κλιματικής αλλαγής αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία της συζήτησης της Κοπενχάγης και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο συνολικός μηχανισμός του χρηματοδοτικού μηχανισμού περιορισμού και προσαρμογής και μοιράσματος του α, ε, βάρους θα αποτελέσει βασικό σημείο της επιτυχίας ή μη των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Συμβούλιο, το καθαρό κόστος προσαρμογής και μείωσης από τις χώρες θα μπορούσε να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ κατ' μέχρι το 2020 και αυτό μπορεί να βρεθεί από τη διεθνή αγορά άνθρακα, τις προσπάθειες των ιδιωτικών χώρων και διεθνή δημόσια χρηματοδότηση. Αυτό το τελευταίο υπολογίζεται μεταξύ 22 και 50 δισεκατομμυρίων ευρώ το έτος έως το 2020 και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε σημαίνει πως θα πρέπει να μοιράσουμε τα βάρη δίκαια σε παγκόσμιο επίπεδο και να, έχουν, να έχουμε ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο. Τεράστια σημασία βεβαίως έχει το να ξεκινήσουμε γρήγορα τη διεθνή στήριξη του 2010-2013 για να προετοιμαστούμε για αποτελεσματική δράση μέσω μακροπρόθεσμη και όπως ξέρετε αυτή η στήριξη υπολογίζεται μεταξύ 5 και 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τώρα, Ο βασικότερος μηχανισμός χρηματοδότησης είναι βέβαια στα δημόσια οικονομικά και η κυριότερη διαπραγμάτευση στην Κοπενχάγη. Και το ζήτημα είναι ποιος και με ποια κριτήρια θα υπομειστεί αυτό το βάρος και πώς θα γίνει η κατανομή παγκοσμίω. Πρώτη παρατήρηση, το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την κατάσταση ανήκει οπωσδήποτε στον ανεπτυγμένο και στις ανεπτυγμένες και βιομηχανοποιημένες χώρες οπότε πρέπει να αναλάβουν και το κύριο βάρος. Είναι όμως αλήθεια πως και κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες, οι πιο ανεπτυγμένες, παίζουν ε, ένα όλο και μεγαλύτερο ρόλο στις παγκόσμιες εκπομπές, κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραβλεφθεί κατά διάρκεια λήψης των αποφάσεων περιορισμού και ε, του πώς θα μοιραστούμε το βάρος αυτό. Χρειάζεται λοιπόν πολιτική θέληση και από τις αναψώμενες χώρες, αλλά και φιλόδοξες δεσμεύσεις από τις ανεπτυγμένες χώρες. Συνολικά, η βοήθεια στις αναψώμενες χώρες για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις μέσω τη οικονομική στήριξη τεχνολογία και μεταφορά τεχνογνωσία θα είναι προ το συμφέρον μα, καθώ θα περιορίσει τι αρνητικέ ε, κοινωνικές αλλαγές όπως οι εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων, πολλαπλασιασμό των περιφερειακών συγκρούσεων λόγω περιορισμού των φυσικών πόρων, επιδείνωση των κοινωνικών ανισοτήτων και της παγκόσμιας στόχης. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιμείνει στην δέσμευσή της να αναλάβει ένα, το κομμάτι εκείνο που της αναλογεί από το κόστος και να ζητήσει και από άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο χωρίς να υποβαθμίσει την καταπολέμηση της στόχιας και τη συνεχή πρόοδο προς τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Δεύτερη παρατήρηση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ε, οικονομικές ε, συνέπειες κλιματικής αλλαγής που θεωρούνται από κάποιους εμπόδιο στην ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Π.χ. δράσεις για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου μοιάζουν κάτι το επικίνδυνο όταν υπάρχει μείωση της βιομηχανικής παραγωγής, κάτι το ακριβό για τον βιομηχανικό κλάδο στην Ευρώπη και με υψηλό κόστος για τις εθνικές οικονομίες. Σας μείνουμε όμως τα νούμερα. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, το ετήσιο κόστος προβλεπόμενης κλιματικής αλλαγής θα είναι μεταξύ 5 και 20% του ΑΕΠ του 2050, ενώ οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν εάν, ξεκινώντας από σήμερα, 1% του ΑΕΠ αφιερώνεται κάθε χρόνο σε μέτρα στον κλάδο αυτόν, όπως αναφέρει η έκθεση Florence. Επιπλέον, είναι σαφές πως έχει διαφορετικές πτυχές η κρίση που αντιμετωπίζουμε, οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές που σχετίζονται με το παρόν μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται σε, διαφορετικό, σε διαφορετικές ανισότητες. Οπότε το να επιστρέψουμε στην κατάσταση προ της οικονομικής κρίσης, το πρώτερο καθεστώς, δεν θα πρέπει να θεωρείται η λύση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι η πολλαπλή αυτή κρίση να μεταβληθεί σε μια ευκαιρία να περάσουμε σε ένα άλλο οικονομικό μοντέλο όπου η αηφορία είναι η λέξη κλειδί. Αηφορία όχι μόνο των φυσικών πόρων, αλλά και μιας οικονομίας χαμηλού άνθρακα όλων των κλάδων της παραγωγής, αηφορία της αγοράς με νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και προώθηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, αηφορία της εργασίας και αηφορία της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οπότε το να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να τη χρηματοδοτήσουμε είναι πολύ περισσότερο από περιβαλλοντική πολιτική. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να στραφούμε σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα προσφέρει ευκαιρίες για τις μελλοντικέ γενιές και θα δημιουργήσει ε, βιώσιμες συνθήκες ζωής για το μέλλον αντί στο να ε, εστιάζουμε το πώς θα διαφυλάξουμε δουλειές και επιχειρήσεις μόνο για σήμερα. Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Εκεί πέρα πρέπει να δείξει το δρόμο η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ψάξει συμμαχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα μπορούμε αμέσως να περάσουμε στην κυρία Κλάδα. είναι η πρώτη μας ομιλήτρια, η κυρία Μακλέτ. Σα ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σα ευχαριστώ που μου δίνετε απόψε την ευκαιρία να σα απευθύνω το λόγο. Εγώ λοιπόν δεδομένη τη τόσο ωραία συναρτήρια ομιλία, δεν θα σα κουράσω με τι λεπτομέρειε των διαπραγματεύσεων και το που βρισκόμαστε αλλά θα ήθελα απλά να πω ότι και μάλλον να θυμίσω τους στόχους όσον αφορά τις εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου και πώς οι στόχοι μείωσής τους σε όλους τους τομείς θα βοηθήσει ε, τόσο για την Ευρώπη, αλλά όσο και αφορά τη θέση της Ευρώπης σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό που θέλω να σας αναφέρω είναι πώς θα πετύχουμε τους ε, τωρινούς και τους μελλοντικούς στόχους, πώς θα περιορίσουμε το κόστος ε, αυτών όλων για την κοινωνία και ο στόχος δεν είναι μόνο να βρούμε το φθηνότερο τρόπο για να μειώσουμε τις εκπομπές, αλλά να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές μας και οι δράσεις μας παράγουν ε, παράπλευρα ωφέλη ώστε ε, και ίσως και το πιο σημαντικό είναι να μην δημιουργήσουμε και προβλήματα αλλού. Αυτή η αλληλεξάρτηση της πολιτικής με τις επενδύσεις είναι αυτό στο οποίο θέλω να εστιάσω την προσοχή μου. Οπότε στο τέλος θα μιλήσω σε σχέση με το γύρο ε, των, οικονομικών επενδύσεων και τις πολιτικές εδώ στην Ευρώπη σε σχέση με το κόστος της προσαρμογής και του περιορισμού, καθώς και τα θέματα που θα μπορούσαμε να μας βοηθήσουν να περιορίσουμε το κόστος και τους κινδύνους. Επίσης θα μιλήσω για την έξυπνη υποδομές και την οικονομία της ε, γνώσης. Δύο πράγματα για τα οποία ιδιαίτερα προσπαθούμε στο δικό μου οργανισμό και θέλουμε τουλάχιστον να διατυπώσουμε κάποιες προτάσεις. Και τέλος, επειδή μόλις έφτασα από το Πεκίνο μετά από πολύ έντονες διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις στρατηγικές του ελέγχου για τον άνθρακα και τις σχετικές επενδύσεις, να σας ενημερώσω για το τι συμβαίνει εκεί, γιατί είναι πιστεύω πολύ σημαντικό καθώς θα πάμε στην Κοπεχάγη. Εγώ δεν χρειάζεται να σας ανακεφαλαιώσω με αριθμούς. Ε, τα γνωρίζετε τα στοιχεία. Είμαστε πάντως σε μια τροχία που μας φέρνει κοντά στο στόχο των δύο βαθμών και γι' αυτό και προβλέπουμε ότι οι παγκόσμιες εκπομπές θα φτάσουν σε μια εχμή το 2020. Να σας θυμίσω ότι το 2020 είναι ε, ο στόχος του Κιώτο, αλλά εκτός από την συμφωνία του, τη δική μας, ε, κανένας άλλος δεν έχει δεσμευτεί αυτή, άρα λοιπόν θα πρέπει να ασκήσουμε την ε, δύναμη επιθούς που έχουμε. Ε, θα πρέπει να φτάσουμε ε, κάτω από τα επίπεδα του, του 1990 μέχρι το 2050, αλλά αυτό το στόχο θα πρέπει να τον, να τον αναλάβουν οι ανεπτυγμένες χώρες και να περιορίσουν τις εκπομπές τους στο 80-95% μέχρι το 2050. Αυτό ε, τονίστηκε και από τους G8 στην Άγκουιλα. Ε, εάν το καταφέρουμε αυτό, θα αν θέλουμε να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να περιορίσουμε τις εκπομπές σε 6% ετησίως, γιατί διαφορετικά μπορεί να αγγίξουμε κάποια πλανητικά κατόφλια. Αυτά είναι πραγματικά δεν είναι κάτι το οποίο συζητείται μόνο στο ίντερνετ, είναι κάτι που θα συμβεί οπωσδήποτε. Και η φιλοδοξία που είχαμε μέσω του πρωτοκόλλου του Κιώτο, που ήταν λιγότερο από τα 6% για ένα μέρος των συμπογραφώντων και μια δικατία για να το επιτύχουμε, αυτό θα πρέπει να το προσπαθούμε και να το επιτυγχάνουμε ετησίως. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Στέν, θα, όπως είπε και ο κύριος Στέν, είναι ε, τώρα η κατάλληλη στιγμή να δράσουμε. Τώρα, οι προσπάθειες που κάνουμε για, στο πακέτο μας CARE για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια είναι πολύ σημαντικές και έχουν τεράστιο αντίκτυπο για την πολιτική για τη ρήπανση της ατμόσφαιρας και θα μιλήσω και για τα παράπλευρα ωφέλη. Με βάση την ανάλυση μας ε, στην ε, οργανισμό μας για ε, τις μεταφορές, τη γεωργία, την ενέργεια και άλλους τομείς, αν εφαρμόσουμε τις πολιτικές υπό το πακέτο CARE αποτελεσματικά, θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε την Ευρώπη σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, θα αυξήσουμε την ασφάλεια ενέργειας, θα ενθαρρύνουμε, πιστεύω, την καινοτομία και νέες ευκαιρίες επιχειρηματικές, καθώς και θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Σήμερα είχαμε επαφή με τον πρόεδρο της που είπε είπε ότι μάλλον είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που είχαμε ποτέ μπροστά μας και αυτό το υπολογίζω όταν, ε, όταν ο κύριος Στέρν είπε το αντίθετο, ότι δηλαδή οι κλιματικές αλλαγές είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της αγοράς μέχρι στιγμής. Δεν θα μιλήσω λοιπόν για τους δεσμευτικούς στόχους, φαντάζομαι τους γνωρίζετε. Ε, την αναλογικότητα που θα έχουμε αν φτάσουμε σε συμφωνία στην Κοπενχάγη σε σχέση με το τι θα είναι οι στόχοι μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου για την ανταλλαγή, μάλλον την εμπορία εκπομπών, αλλά και εκτός αυτού. Ήμουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος πριν από μία εβδομάδα και μου ετέθησαν πολλές ερωτήσεις από νέους βουλευτές και κάποιους σκεπτικιστές και κάποιους που δεν πιστεύουν και πολύ τα στοιχεία, αλλά θα σας διαβεβαιώσω πως η Ευρώπη έχει μειώσει τις εκπομπές της. Είμαστε ε, εντάξει με τους στόχους μας ε, του Κιώτου και αν βάλουμε τις εκπομπές των 27 είμαστε 10% χαμηλότερα το 2008 από το 1990. Μετά από το τέταρτο έτος λοιπόν της προσπάθειας έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τους στόχους και δεν είναι αυτό αποτέλεσμα μόνο της ύφεσης ή των οικονομικών επιπτώσεων αυτής. Έχουν τεθεί φιλόδοξοι στόχοι για την ανανεώσιμη ενέργεια. Η Φιλανδία, η Σουηδία και η Αυστρία πετυχάνουν στόχους που ήταν πολύ πιο πέρα από τους ε, προσυμπεφωνημένους. Πολλές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούν να φτιάξουν νομοσχέδια φιλόδοξα που θα μας οδηγήσουν στα μέσα του αιώνα σε περιορισμούς ε, των εκπομπών ε, των αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 με 95%. Αυτό σημαίνει 10 τόνους εκπομπές έχουμε αυτή τη στιγμή ε, διοξιδίου του άνθρακα ετησίως. Κατά κεφαλήν θα πρέπει αυτό να περιοριστεί στους 2 τόνους. Αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να το προβλέψουμε με τρόπο που να έχει αποτέλεσμα. Στα τελευταία 30 χρόνια έχουμε περάσει πάνω από 100 δις για, την, για γεγονότα που σχετίζονταν με την ξηρασία και ε, οι αριθμοί συνεχίζουν να αυξάνονται. Βλέπουμε λοιπόν ε, σχετικές ζημιές, βλάβες και σίγουρα τα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι καλύτερα. Και το χειρότερο είναι γύρω από την Μεσόγειο και έχουμε κάνει και σχετική έκθεση για τις Άλπεις. Ο τομέας των μεταφορών ε, αρχίζει να βρίσκει ανομαλίες για το κατά πόσο τα πρόσφατα, οι πρόσφατες πιλωτικές έρευνες δείχνουν δραστικές πτώσεις στις ε, θερμοκρασίες. Ορισμένε φορές ε, μείον 70 έχουν φτάσει στις θερμοκρασίες σε σημεία όπου δεν είχαν παρατηρηθεί τέτοιου είδους θερμοκρασία. Εκραία γεγονότα λοιπόν που προκαλούν ε, ζημιές σε παλιές υποδομές. Γενικά λοιπόν οι κλιματικές αλλαγές θα μας υποχρεώσουν να διαρθρώσουμε πολλά από αυτά που κάνουμε και ε, κάτι το οποίο σύμπτωμα θα πρέπει να σας απασχολήσει είναι η εξάρτησή μας από πρώτες ύλες. Είμαστε σαφώς σε ανταγωνισμό με την Κίνα και την Ινδία, ιδιαίτερα για την αυξανόμενη ζήτηση πόρων. Η Ευρώπη σαφώς δεν, ε, ε, μάλλον είναι παραγωγός και κατασκευαστής, όμως ε, οι ελλείψεις στην κατασκευή και στην μεταποίηση θα απαιτήσουν θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία μας. Δηλαδή διαφορετικούς πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την παραγωγή ενέργειας, λύσεις σε πιο πιο αποτελεσματικές για τις μεταφορές, για τις πόλεις κτλ. λοιπά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μόλις ολοκληρώσαμε μια έκθεση από το Διεθνές Πάνελ της UNEP για την βιώσιμη χρήση των πόρων και εξετάζουμε εκεί τα μέταλλα. Τέσσερα είδη μετάλλων, τα σιδηρούχα, τα μη σιδηρούχα, αλλά εμένα με ενδιαφέρουν περισσότερα τα, τα πολύτιμα μέταλλα. Αυτά το αντιμόνιο, μόλιβδος και, που, εξα, που εξορίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό αλλά και ανακυκλώνονται. Αυτά είναι τα μέταλλα τα οποία στα οποία βασίζεται η σύγχρονη μας ε, κοινωνία. Είναι αυτά που υπάρχουν στα τηλέφωνα, στα διάφορα καλώδια που περνούν από όλη την Ευρώπη. Είναι τα νέα υλικά που βλέπουμε στις ε, στα αυτοκίνητα και στα αεροπλάνα. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι οι σχέσεις γονιού με θυγατέρα σε αυτά τα υλικά, όπως ξέραμε για το χαλκό, για το αλουμίνιο κτλ. Βασιζόμαστε ε, πάρα πολύ σε αυτή την εξόριξη του μεταλλεύματος για να μας δώσουν αυτά τα στοιχεία σίγουρα όταν δεν απαιτείται τόσο πολύ σχάλιβας για να οικοδομήσουμε ε, τις υποδομές μας, αν δεν έχουμε φτιάξει καλή ανακύκλωση για αυτά τα υλικά, διατρέχουμε τον κίνδυνο να έχουμε έλλειψη σε κάποιες από τις πιο καινοτόμες ε, προτάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να επιστιάσουμε την προσοχή μας στην ανακύκλωση αυτών των πρώτων υλών. Επίσης, ε, βιοκαύσιμα. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι κάποιες σοφές αλόγιστα ίσως ε, παρουσιάσαμε το θέμα και αυτή η έκθεση είναι η πιο εμπεριστατωμένη που έχουμε ενώπιον μας και τονίζει το γεγονός ότι τα βιοκαύσιμα έχουν το χώρο τους, αλλά με βάση ορισμένους όρους μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κάνουμε τέτοιου είδους δουλειά θα πρέπει να αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα κάθε επένδυση αλλά και ε, θα πρέπει δηλαδή να προβλέψουμε και τις ε, επενδύσεις ως αντίβαρο που θα πρέπει να γίνουν αν δεν λειτουργήσει το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την, απο, την αποτελεσματικότητα για να μπορέσουμε στα επόμενα χρόνια να, να, να πετύχουμε τους στόχους. Η McKinsey ε, εκτιμά πως χρειαζόμαστε 30 δις ευρώ ετησίως να δαπανώνται για την επάρκεια ενέργειας με βάση τις υπάρχουσες τεχνολογίες για να βασιστούμε δηλαδή 10% ή περισσότερο στις επενδύσεις. Και έτσι φτάνουμε στους στόχους μας για το 2020. Ε, τονίζουν λοιπόν τον χώρο που έχουμε θετική ε, ε, κέρδος για τις επενδύσεις και σε ολόκληρο τον κόσμο η πάρκια σε ενέργεια και απόδοση της ενέργειας απασχολεί τον κόσμο. Αν δούμε όμως ε, τα σχέδια ανάκαμψης και μάλιστα υπήρχαν 17 χώρες που έφτιαξαν ως τμήμα των πράσινων μέτρων τους τέτοια μέτρα, τα ποσά που δαπανώνται για την επάρκειας ενέργεια είναι σχετικά μικρά. Μιλάμε για επάρκεια ενέργειας, ανανεώσιμες ενέργειες, ε, για την ε, διάλυση αυτοκινήτων, προγράμματα υδροδότησης κτλ. Αυτά είναι μέτρα που, αφορούν, που περιλαμβάνονται στα οικονομικά πακέτα. Όμως είναι σαφέ πω τα χρήματα αυτά σε ορισμένε περιπτώσεις δεν είχαν τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν αν είχαν συνδυαστεί με άλλου είδου πολιτικές, όπως για παράδειγμα αυτές που φορούν τα κτίρια. Χρειάζονται λοιπόν να στοχευθούν τα μέτρα με θετικές και αρνητικές αναλύσεις και αν το κάνουμε αυτό μπορούμε όντως, όπως είπε και η Αντιπρόεδρος, να αποφύγουμε τον αντίκτυπο των κλιματικών αλλαγών μέχρι και 50% ε, του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αυτό θα πρέπει να κινητοποιήσει τις καινοτομίε, την ασφάλεια σε ενέργεια, όπου μπορεί δυνητικά να δούμε τον περιορισμό φυσικού αερίου ή και πετρελαίου κατά 50% ετησίως. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι περιορίζεται η ανάγκη κατά 11 δις για λήψη μέτρων για την ε, ρήπανση του αέρα. Αυτά ισχύοντα για την ρήπανση του αέρα έχουν ως αποτέλεσμα κέρδος ε, της τάξης των 64 δις όσον αφορά τα υγειονομικά έξοδα που θα είχαμε αν δεν είχαμε λάβει τα μέτρα αυτά. Να στραφώ λοιπόν ε, ε, γρήγορα στην Κίνα. Η Κίνα προσπαθεί να ελέγξει τη χρήση του άνθρακα, κλείνει τις ε, ρηπογόνες εταιρείες, περίπου 700 από, από τις μικρότερες τους εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σκοπεύουν να, να τις τα κλείσουν μέχρι στα επόμενα χρόνια και επίσης 700 ε, εκατομμύρια ευρώ προσφέρουν για τα, ως ανταμοιβή για τα πιο οικονομικά σε ενέργεια προγράμματα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι στο πακέτο του, στο 40% είναι ειδικά με πράσινο προφίλ, αλλά το 38% αφορά τις υποδομές, ε, σιδηροδρόμους έχουν το μεγαλύτερο δίκτυο ε, ταχύων σιδηροδρόμων στον κόσμο. Ε, έχουν ε, είναι η μεγαλύτερη παραγωγή σε αιωλική ενέργεια και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα κρίσιμο ε, πρόγραμμα το οποίο φτιάχνουν, ε, εμείς δεν το έχουμε, αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι πως κάθε μέτρο πολιτικής και κάθε επένδυση που κάνουν βλέπουν τα ε, παράπλευρα ωφέλη σε σχέση με την ρήπανση του αέρα, το νερό, την πρόσβαση στο νερό. καθημερινή του ζωή λοιπόν έχει μετατραπεί ώστε να συνδυάζονται αυτές οι πολιτικές σε κάθε βήμα αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και είδα τα στοιχεία αυτό το Σαββατοκύριακο ότι θα επιτύχουν τους δικούς τους στόχους για μείωση της, των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου ε, μέχρι το 2020 και ίσως και λίγο παραπάνω από τους ε, στόχους που είχαν θέσει. Τέλος υπάρχουν ένα περισσότερο, υπάρχει όλο ένα περισσότερο ζήτηση για γνώση. Υπάρχουν όλο ένα περισσότερο γνώσεις και είναι πολύ ενδιαφέρον που βλέπουμε ότι οι εταιρείε είναι πρόθυμες να προσφέρουν τα στοιχεία τους για να δούμε, να βελτιώσουν μάλλον τις δικές μας γνώσεις για το πόσο αποτελεσματικές είναι οι πολιτικές μας. Ε, Οποιαδήποτε από τι εταιρείε με τι οποίε εμεί έχουμε να κάνουμε είναι πολύ πέρα από αυτά τα συγκεκριμένα πακέτα ή τα ποσά που έχουν να προταθεί από τι εθνικέ κυβερνήσει. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι είναι, ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα σε όλα αυτά. Η πρότασή μα είναι να εξετάσουμε προγράμματα που θα μα δώσουν περισσότερε στοιχεία και πληροφορίε για να δούμε πώ μπορεί να προκύψουν τα διάφορα παράπλευρα ωφέλη και νομίζω πως αυτό είναι το πιο θετικό στοιχείο που προκύπτει από το πακέτο CARE. Ένα πρόγραμμα υπάρχει το Παγκόσμιο Πρόγραμμα για την, περιβάλλον, για την Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και την Ασφάλεια είναι ένα από τα προγράμματα για τα οποία είναι αρμόδια δική σας Επιτροπή. Είναι ένα ε, διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα και αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τους συναδέλφους της ΕΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά αυτό που σίγουρα κάνει και είμαι ευτυχής ότι ένα-δυο μέρες θα το ξεκινήσουμε, ότι συγκεντρώνει τις πληροφορίες που έχουμε, πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει εδώ και πολλά χρόνια, τα θέτει στη διάθεση των πολιτών και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων με τρόπο που να έχει νόημα για τις καθημερινές του δράσεις. Πιστεύω πως το GMS θα το κάνει αυτό για τις βιομηχανίες. Ήδη προετοιμάζουμε υπηρεσίες κλιμα... κλιματολογικές. Θα κρατήσει αυτό ασφαλή ε, τα αεροπλάνα στον ουρανό, τα πλοία αλλά και τα τρένα και θα μας πει πολλά για το πού ακριβώς οι κλιματικές αλλαγές μας καθιστούν ε, ευάλωτους. Εγώ σας το συστήνω λοιπόν, ελπίζω πως ε, στα επόμενα δύο χρόνια θα μπορέσουμε να δούμε πώς αυτές οι επενδύσεις ως ένα δημόσιο αγαθό μπορούν να μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα με πολύ ψηλή ποιότητα ε, περιβάλλοντος και ζωής για τους ανθρώπους που ζουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Για να μην χρονοτριβούμε, μπορούμε να περάσουμε μέσα στον επόμενο εμπειρογνώμονα μας. Ε, είχαμε καλέσει τον Νίκολα Σέρν, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι παρόν και μας έχει στείλει ένα μήνυμα βίντεο. Παρακαλώ να μας το παρουσιάσετε. Ελπίζω να λειτουργήσει η τεχνολογία. Για να ακούσουμε την άποψη και του κύριου Stern, του Λόρδου Stern. Ένα λεπτό, να αρχίσει. Hello, my name is Nick. Καλημέρα σας, λέγομαι Nick Stern και σας μιλάω από το London School of Economics. Yeah, to have extensive discussions on India's climate change action plans, and that's why I can't be with you.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 Ο επόμενο μιλήσει ο κύριο Κούμαρ. Σα καλωσορίζω. Και σα δίνω το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Χέρμπερτ Ρόιλ, κυρία Ποδηματά, συνεπειρογνώμονες, αγαπητοί επισκέπτες, κατά βάση θα αναφερθώ πάνω σε κάποια αποτελέσματα που ίσως έχουν επιπτώσεις στις κτηματολογικές αλλαγές. Ε, αποτελέσματα αυτό. Τι μπει, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Που αφορά την οικονομία της βιοπικυρομορφίας και η μελέτη αυτή θα ολοκληρωθεί το 2010, αλλά έχουμε κάποια προσωρινά αποτελέσματα που μπορούμε να παρουσιάσουμε και θα περιοριστώ σε εκείνα τα αποτελέσματα που έχουν πραγματικά επιπτώσεις στις κλιματολογικές αλλαγές. can move further. See, so basically, three findings I would like to... Κατά βάση υπάρχουν τρία αποτελέσματα που θα θέλω να σας παρουσιάσω. Το πρώτο είναι η δημιουργία των κορολογιανών ε, υφάλων και προβλέπεται ότι λόγω των κλιματολογικών αλλαγών αυτό, αυτοί οι κορονογενεί ύφεδοι απειλούνται. Και τι θα χάσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται αυτό που το TIP έχει αυτά τα αποτελέσματα αλλά πρώτη φορά συζητιέται όχι μόνο για την φυσική καταστροφή, αλλά και για τις επιπτώσεις που θα μπορεί να έχει η απώλεια αυτών των κοροϊδικών υφάλων. Το δεύτερο θέμα είναι οι αλλαγές μέσω του πράσινου άνθρακα. Θα σας πω τι είναι ο πράσινος άνθρακας. Και το τρίτο είναι η προσαρμογή με την επαναφορά των οικολογικών συστημάτων. Αυτά είναι. Λοιπόν, όπως ξέρετε, το TIP είναι από την Κομισιόν, την την ΤΕΦΡΑ, και το Γερμανικό Αρμόδιο Υπουργείο, το Νορβηγικό, το Ολλανδικό και άλλα. Η προσελνή έκθεση που παρουσιάστηκε πέρσι είχε τρία βασικά αποτελέσματα. Το πρώτο ήταν το πώς λόγω των απολειών στα οικοσυστήματα μειώνεται η ευμάρεια των πολιτών. Υπάρχουν μάλιστα κάποια στοιχεία που λένε ότι οι απώλειες αυτές είναι της τάξη του 6-7% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Ίσως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά οι απώλειες αυτές οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το δεύτερο αποτέλεσμα που υπάρχει στην προσωρινή αυτή έκθεση δίνει την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο οι απώλειες του MDG που θα ε, ε, αυξηθούν με την πλήξη στα οικοσυστήματα, αλλά και όλοι οι άλλοι δείκτες θα μειωθούν σημαντικά λόγω της μείωσης στην ε, βιοπικερμορφία και την επιδείνωση κατάσταση των οικοσυστημάτων. Το τρίτο αποτέλεσμα είναι πώς θα επιλέξουμε τους παράγοντες ε, μείωση της τιμής και πώς θα μπορεί οι μειώσεις αυτές να είναι τελικά ηθικής μορφής επιλογές. Αυτό είναι η προσωρινή έκθεση. Και θα σας δώσω κάποια ιδέα για τη δομή της έκθεσης. Υπάρχουν πέντε κύριοι παράγοντες που είναι στοχευμένοι σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές. Δηλαδή επιστήμονες, η ε, πολιτική, η διοικητική, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες και καταναλωτές. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα πλαίσιο που αποκαλείται D0 Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι το πλαίσιο για το τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ μπορείτε να δείτε ότι εδώ έχουμε το D1, D2, D3 και D4 αλλά την επιστημονικά, τα επιστημονικά στοιχεία προέρχονται από το D0, D0. Αυτό τι σημαίνει για τις κλιματολογικές αλλαγές ε, σύμφωνα με το TIP. Καταρχήν, όπως σας είπαμε, το θέμα των κολογεγονών υφάλων. Και αυτό προήρθε από μια ενημέρωση των κλιματολογικών αλλαγών και που θα παρουσιαστεί κατά πάσα πιθανότητα στη διάσκεψη της Κοπενχάγης τον επόμενο μήνα. Όπως βλέπετε, τα κοράλια ε, που υπάρχουν σε κρύα ψυχρά ύδατα και σε θερμά ύδατα κατανέμονται με αυτόν τον τρόπο που είδατε στο χάρτη. Και υπάρχουν διάφοροι τύποι αποτελεσμάτων ανάλογα με την αξιολόγηση που γίνεται. Ότι περίπου το 30% των κορολογιανών υφαλών απειλούνται. Αυτό τι σημαίνει όσον αφορά τις οικονομικές απώλειες. Προσπαθούμε να δούμε τα στοιχεία και να κάνουμε εις βάθος ανάλυση. Να δούμε γιατί αξίες συζητάμε. Βλέπετε να δείτε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Αν δεν τα βλέπετε καλά, να πάρετε το γραπτό κείμενο στα χέρια σας, παρακαλώ. «83 μελέτες έγιναν που και συνέλεξαν στοιχεία και για τα ψυχρά ε, ύδατα και για τα θερμά ύδατα όπου υπάρχουν τα κοράλια. Το κόστος είναι 4,5 αμερικανικά δολάρια ανά εκτάριο. Αυτά ήταν τα στοιχεία για το 2007. Αυτή ήταν η τιμή. Και προσπαθήσαμε να καταμετρήσουμε τις απώλειες ή τα ωφέλη στα οποία οδηγούμεθα. Απώλειες απώλειες και ωφέλη είναι το ίδιο. Δηλαδή ένα όφελος αποκλείει μία απώλεια και μία απώλεια αποκλείει ένα όφελος. 370 ε, αμερικανικά δολάρια λοιπόν είχαμε ε, κατά μέσο όρο για τις διακανονιστικές υπηρεσίες ήταν 648 δολάρια. Έχετε όμως κάποια ένδειξη του πού είναι οι απώλειες και ποιο είναι το έμβρος των απώλειων αυτών. Και οι πολιτιστικές υπηρεσίες που προέρχονται από την απώλεια των κοραλιών είναι 7.325 δολάρια ανά εκτάριο και έτος και πάντα με τιμές του 2007. Κοιτάξτε, πολλοί ίσως θεωρούν ότι τα κοράλια σε πολλά μέρη του κόσμου έχουν αυτή την εικόνα. Πραγματικά όμως είναι έτσι. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι, διαφορετικές, οι διάφορες κλιματολογικές αλλαγές έχουν επιπτώσεις σημαντικές. Λοιπόν, τα τροπικά κορολογιανή, η τροπική κορολογιανοί υφαλοί βρίσκονται σε μια κατάσταση στην οποία οι απώλειες, η καταστροφή τους δεν θα μπορεί πια να αντιστραφεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και καμιά φορά αυτές οι αναπέτρεπτες ε, αλλαγές σημαίνουν ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Πρέπει να είμαστε σαφείς γι' αυτό. Και άμα μιλάμε για κλιματολογικές αλλαγές, βλέπουμε ότι ό,τι και να κάνουμε δεν θα μπορέσουμε κατά πόσο, πάσα πιθανότητα να α, κερδίσουμε πάλι τα κοράλια αυτά. Τώρα, η ηθική επιλογή είναι σταθεροποίηση στα 450 ppm ή στα 350 ppm του διοξιδίου του άνθρακα. Και αν δούμε την ανάγκη επιβίωσης των ε, τροπικών κοροϊνών υφάλων, είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθήσουμε το 350 ppm και αυτό ε, μας επαναφέρει σε αυτό που είπε ο Σερ Νίκολα Στέρν προηγουμένως όσον αφορά την μείωση και για τις αναπτυσσόμενες αναπτυγμένες ε, ε, ε, περιφέρειες. So in New Delhi, the environmental... Ε, τελευταία, ακούσαμε τους ε, υπουργούς να λένε ξεχάσε το πρωτόκολλο του Μποκ». Εμείς ε, είμαστε φτωχοί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Α, αλλά οι πρωθυπουργοί είπαν ότι εντάξει θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί αυτό το οφείλουμε στις μελλοντικέ γενιές. Λοιπόν, αν θέλει κανένας αυτά 450 parts per million με ανά εκατομμύριο διοξείδιο του άνθρακα, τι πρέπει να γίνει. Να, εδώ έχετε κάποια αποτελέσματα. σήμερα ε, τι γίνεται και ανάλογα με το, τις διαφορετικές οδούς που μπορεί να ε, ακολουθήσει η κλιματολογική αλλαγή έχουμε διαφορετικά σενάρια. Εδώ έχουμε δύο βαθμούς αύξησης θερμοκρασίας, τρεις βαθμούς και βλέπετε πώς μετατρέπονται αυτά τα κοράλια. Αυτό είναι ένα σενάριο και γι' αυτό χρειάζεται κατεπίγουσα δράση για να αποφύγουμε την απώλεια των κοραλιών αυτών. Μετά, το ο άνθρακας από τα δάση για τις κλιματολογικές αλλαγές. Mm-hmm. Different land use Διαφορετικές χρήσεις της γης οδηγούν σε στόχους ε, διοξείδου του ανθρώπου 450 ppm με κοινό φόρο πάνω στις ε, κομπές αυτές. Εάν έχουμε όμως μια διαφοροποίηση, πάλι μπορούμε να έχουμε μεγιστοποίηση του κοινωνικού ωφέλους. Αυτό είναι το μήνυμα από αυτό το διάγραμμα. Άμα έχετε ερώτηση, μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω αποθήκευση ενός τετάρτου όλου του επιγείου άνθρακα και συλλογή μέχρι 4,8 γιγατόνων διοξιδίου του άνθρακα ετησίως. Μπορεί να γίνει όλο αυτό στα δάση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα δηλαδή αυτό από την αξιολόγηση του ΤΥΜΠ. Το άλλο είναι το θέμα της προσαρμογής. Δεν το συζητήσαμε. Προφανώς θα πρέπει να σταθεροποιηθούν οι εκπομπές ε, άνθρακα και να μειωθούν. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, πώς θα μεταφραστεί σε μία προσαρμογή, είναι επίσης σημαντικό και πάνω σε αυτό θα πω δύο λόγια. Αν θέλετε η στρατηγική προσαρμογή να είναι αποτελεσματική, τότε η διατήρηση και επαναφορά των δασών των λιμνών και των υγροτόπων είναι ουσιαστικότητα της σημασίας. Αυτό έχει πολλά οικονομικά ωφέλη, θα σας πω και άλλα πάνω σε αυτά, αλλά αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που απορρέουν από τις έρευνες του ΤΥΠ. Δεύτερον, η παραγωγικότητα της γεωργίας και της αλίας, γιατί τα δάση για τα, τις διάφορες ουσίες και οι ροές των υδάτων θα μπορούσαν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν σαν δυνατότητα όχι μόνο για την προσαρμογή και για τη σταθεροποίηση, αλλά και για την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων. Εάν κάποια κοινωνία, παραδείγματος χάρη, η Κίνα, η Ινδία, η Ινδία έχει ήδη 350 εκατομμύρια φτωχών, αν βασιστεί κανένα με, στη βάση του ενός δολαρίου ανά ημέρα, αν πάμε στα δύο, έχει τα διπλάσια. Ο ημισή είναι φτωχή. Οι επιλογές λοιπόν δεν έχουν εξατεστεί πάρα πολύ προσεκτικά. Και γι' αυτό χαρικά πάρα πολύ για το μήνυμα του Νίκολα Στέρν ότι σχετίζονται στενά η φτώχεια και η κλιματολογική αλλαγή. Το ένα δεν μπορεί να αλλάξει εάν δεν υποστηρίξουμε το άλλο. Και υπάρχουν οι δυνατότητε ενδιαφερόντων σεναρίων, όπου οι ε, πολιτικές προσαρμογές θα μπορέσουν να βοηθήσουν και στην ε, πάνταξη της φτώχειας. Μετά υπάρχουν οι φυσικές ε, καταστροφές. Ε, Παραδείγματο χάρη είναι λειψιδρία, πλημμύρες ε, που μπορούν να περιοριστούν από την ανάπτυξη των δασών. Όταν κανένας ε, συζητά για την επαναφορά στα παλιά επίπεδα, θα πρέπει να δούμε αυτό τι σημαίνει οικονομικά. Η ΤΥΠ ανέλησε διάφορα οικοσυστήματα όπως βλέπετε εδώ. Και στις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε ότι το ποσοστό επιστροφής ή η σχέση ο κόστος ωφελίας είναι υψηλότερο από ότι οποιοδήποτε παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα συμπληρωματικό κίνητρο να γίνουν επενδύσεις στα οικοσυστήματα που όχι μόνο θα μειώσουν το άνθρακα, αλλά θα είναι και καλή επένδυση για τα χρήματά σας. Και υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες αναλύσεων μέσος όρος, ε, οικονομικές τιμές κλπ. Και σε όλες τις αναλύσεις είδαμε ότι είναι απόλυτα λογικό να επενδύσουμε στην ε, πανόρθωση των οικοσυστημάτων. Δύο λεπτά ακόμα και μετά θα κλείσω. Έχουμε ε, καφέ άνθρακα, ε, πράσινο άνθρακα και μπλε άνθρακα. Και βλέπετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να δώσουμε τις σωστές προτεραιότητες στην αποθήκευση του, ε, του άνθρακα και υπάρχει πράσινος ε, γαλάζιος και μαύρος μάλιστα. Και τέλος, τρία μηνύματα που θέλω να συμμεριστώ μαζί σας. Το πράσινο, ο πράσινος άνθρακας δεν είναι εναλλακτική, είναι αναγκαιότητα. θα ήταν απαραίτητο να έχουμε τουλάχιστον το 30% πράσινου άνθρακα. Και τέλος, η επαναφορά, δηλαδή η επαναφορά των οικολογικών συστημάτων είναι εύκολο να ελέγχεται και βλέπετε από την ανάλυση κόστος ωφελίας ότι είναι πολύ ωραία τα αποτελέσματα, είναι πολύ συγκεκριμένα στη στοποθεσία τους, στη γινό και αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος που πρέπει να ακολουθεί η στρατηγική προσαρμογής και για καλές επενδύσεις με καλά αποτελέσματα. Αυτά τα τρία σημεία θα ήθελα να έχετε κατά νου σαν τελευταίο μου μήνυμα. Και θα ήμουν πολύ ευχαρίστω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Herzlichen Dank. Sofort weiter. Die nächste Redner ist Mr. Campbell. Uh, you want to come there. It's better. Mr. Campbell, θέλετε να επανέλθετε. Alle. Σας παρακαλώ όλους να προετοιμαστείτε όταν θέλετε να θέσετε ερωτήσεις ή να παρεμβείτε. Να βιαστείτε λίγο γιατί 5 η ώρα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το ξαναλέω. Οπότε έχουμε καθυστερήσει λίγο. Ο κύριος Κάμπελ τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Και αν έχετε ερωτήσεις, ε, νομίζω μπορεί ο καθένας να περιοριστεί σε ένα λεπτάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ την ευκαιρία που μου δίνετε. Νομίζω ακούσαμε το σαφές μήνυμα από εσάς και τη Συμπρόεδρο πριν από λίγο ότι η χρηματοδότηση είναι κρίσιμη για την επιτυχία της Κοπενχάγης. Πριν ε, ξεκινήσω να τονίσω πως οι επιχειρήσεις είχε, είχαν ή ήθελαν να συνεισφέρουν λίγο στην συζήτηση αυτή και προσωπικά ανησυχώ για το ότι ασχολούμαστε μόνο με τα νούμερα. Ξέρω πως βεβαίως αυτά είναι το βασικό, αλλά έχουμε μανία. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω σύντομα σε αυτή την παρουσίαση είναι να κάνω μια πρακτική προσέγγιση και να δούμε αντίστροφα το ζήτημα. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να απαντήσω είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα μέσα τα οποία θα συμφωνήσουμε στην Κόπενχάγη για να έχουμε το μεγαλύτερο όφελο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό το οποίο θα πω είναι αποτέλεσμα πολλών συζητήσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά όχι κάποια κοινή θέση των επιχειρήσεων. Είναι κρίσιμο για το τι θα αποφασιστεί στην Κοπενχάγη, γιατί χρειαζόμαστε να λειτουργήσει η χρηματοδότηση, αν είναι να φτάσουμε στη μείωση που ζήτησε ο κύριος Στέρν, η κυρία Γκλέιτ και η Λυπή. Αυτό θα συμβεί εάν ευθύ εξ αρχής, ενώ δηλαδή από την Κοπενχάγη ήδη, αποκτήσουμε τις κατάλληλες διαδικασίες. Αλλιώς χωρίς αυτούς τους ελέγχους, πολλά από τα χρήματα θα σπαταληθούν και θα χάσουμε μια χρυσή ευκαιρία. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω έχετε τις διαφάνειας, κάποιες φαίνονται, δεν ξέρω αν φαίνονται στην μεγάλη οθόνη. Ε, μπορούμε να αλλάξουμε διαφάνεια. Yes, they are working. So what do I have? To, so which what did I? Okay, the space bar. Okay. Okay, fine. We have sides working down there in a different way from. Ωραία εσεί βλέπετε άλλε διαφάνειες από εμένα, εν πάση περιπτώσει θα αυτοσχεδιάσω. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στην διπλή πρόκληση στον τομέα της ενέργειας. Πρώτα απ' όλα, να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και στην καλύτερη πρόσβαση στην ενέργεια και δεύτερον στον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής. Εάν τα θέσουμε σε ένα πλαίσιο, βλέπουμε από την ε, Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, μιλάμε 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην ενέργεια, 45-3 εκατομμύρια δολάρια θα χρειαστούν μέχρι το 2030 για τους κινδύνους από το κλίμα. Οπότε πρέπει να φτάσουμε σε επιταχυμένη ανάπτυξη και χρήση υπαρχουσών και προηγμένων τεχνολογιών που εκπέμπουν λίγα αέρια του θερμοκηπίου, εάν είναι να επιτύχουμε τις φιλοδοξίες μας με ένα κόστος το οποίο μπορούμε να πληρώσουμε. Ας δούμε λοιπόν τα βασικά μας αυτά, τις βασικές σκέψεις στον τομέα της χρηματοδότησης. Κλίμακα και προβλεψιμότητα. Αυτό το ακούμε σε κάθε συνεδρίαση. Καλά είναι να μιλάμε για τα νούμερα, χρειαζόμαστε προβλέψιμότητα. Δηλαδή να έχουμε ένα προγραμματισμό για σειρά ετών. Κατόπιν, πηγές από πού θα έρθουν αυτά. Πώς θα διακυβερνηθούν. Στόχος και επιλεξιμότητα. Και τέλος το ότι πρέπει να είναι διαρκής η χρηματοδότηση. Εάν δούμε λοιπόν το μέγεθος Μιλάμε για μεγάλα νούμερα, 100 δισεκατομμύρια το έτος τουλάχιστον. Μιλάμε για υψηλά μεγέθη. Όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, τα χρήματα θα είναι δημόσια και ιδιωτικά από τις αγορές και τις αγορές, τα χρηματιστήρια του άνθρακα και βεβαίως ε, μιλάμε για διαφανείς ε, κανόνες, ανοιχτή επιλεξιμότητα και σαφείς απαιτήσει. Θα επανέλθω εδώ πέρα και τέλος μιλάμε για μεγάλες ροές πλούτου και επενδυτικές. Και είναι σοβαρό αυτό. Δεν είναι μικρό θέμα. Εάν δούμε λοιπόν τις συζητήσεις που είχαμε, νομίζω πως μία από τις ε, βασικές πτυχές είναι πως θα πρέπει να προωθηθεί και να μοχλευτεί η ιδιωτική επένδυση όπως υπόθηκε εντός και εκτός του ζητήματος κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να γνωρίζουμε πως τα προηγούμενα που θα δημιουργήσουμε τώρα μπορούν να μας βοηθήσουν αλλά και να μας εμποδίσουν στο μέλλον όσον αφορά την πρόοδο. Κάτι το οποίο βλέπουμε στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο οι επιχειρήσεις ε, θεωρούν ότι πρέπει να προωθηθεί, είναι η ανάγκη αρχικής χρηματοδότησης για να δημιουργηθούν το δυναμικό. Και επανέρχομαι εδώ πέρα, δεν πρέπει να σπαταλήσουμε τα χρήματα που έχουμε, πρέπει να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα. Αλλιώς θα εξαφανιστούν, αν δεν, υπάρχει, λοιπόν, κατάλληλες, αν δεν υπάρχουν κατάλληλες δυνατότητες. Και τέλος μιλάμε πράγματι για α, ανακατανομή πλούτου και πρέπει αυτό να το πουλήσουμε στο κοινό. Βλέπουμε τις παρουσιάσεις για τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής. Ε, έχουμε πείσει το κοινό αρκετά για να καταλάβει το κίνδυνο για να δεχτεί αυτές τις μεταφορές πλούτου. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στη δημόσια χρηματοδότηση και το τι εμείς ε, βλέπουμε ως ρόλο της δημόσιας χρηματοδότησης και ελπίζω τώρα να φαίνονται οι διαφάνειες, νομίζω από την πλευρά των επιχειρήσεων θέλουμε ο πολιτικός και τεχνολογικός κίνδυνος να μειωθεί για να έχουμε και περισσότερη ιδιωτική χρηματοδότηση έργων που αλλιώς δεν θα ήταν βιώσιμα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε πως τεχνολογίες υψηλού κινδύνου να χρηματοδοτηθούν κατά τη φάση επίδειξης και τέλος να κλείσει το κενό μεταξύ των έργων που είναι συνήθι, ας πούμε, και το υψηλότερο κόστος που σημαίνουν οι προχωρημένες τεχνολογίες. Οι εταιρείε έχουν πρόβλημα με το να εξασφαλίσουν κεφάλαια εκ των προτέρων. Εδώ πέρα μπορεί λοιπόν να βοηθήσει η δημόσια χρηματοδότηση για τα έργα τα οποία είναι έντασης ενέργειας και κεφαλαίου. Οπότε Ένα καλό τρόπο βεβαίως να επιβραβεύονται όσοι ε, προσπαθούν να επιτύχουν μια καινοτομία και, και οι ανταμοιβέ του θα πρέπει να είναι βεβαίω προβλέψιμε για να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία καινοτομία και ανάπτυξη των τεχνολογιών και προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια. Εάν λοιπόν δούμε τώρα κάποιες από τι αρχές και είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ ως επιχειρήσεις, μας ανησυχεί πάντα το να δούμε ποιος θα χάσει και ποιος θα κερδίσει και οπωσδήποτε πιστεύουμε πως οτιδήποτε γίνει με δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να είναι ουδέτερο όσον αφορά την τεχνολογία. Οπότε δεν πρέπει να ευνοήσουμε τον έναν παραγωγό μόνο. Έχει συμβεί στο παρελθόν, επικίνδυνο προηγούμενο. Και το έχω αναφέρει και στο παρελθόν, διαφάνεια και προβλεψιμότητα είναι κέρυες, γιατί όταν μια επιχείρηση, τότε η επιχείρηση ξέρει ε, πότε να ζητήσει αυτή την χρηματοδότηση. Και η ισότητα. Δεν έχει σημασία από πού προέρχεται η κοινοτομία, από ποια χώρα, εντός, εκτός Ευρώπης, ανεπτυγμένη χώρα, αναπτυσσόμενη, δεν έχει σημασία πρέπει να διασφαλίσουμε, αν μιλάμε για δημόσια χρηματοδότηση για την καταπολέμηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, πως υπάρχει ισότητα στις ευκαιρίες ανταγωνισμού. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την καινοτομία, να ενθαρρύνουμε τις εταιρείες που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές. Έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, θα συνεχίσουν την καινοτομία και πιθανώς με διαφορετικό τρόπο θα καταλήξουν σε άλλη λύση. Πρέπει να τις ενθαρρύνουμε. Και πάλι πρέπει τα χρήματα να είναι αρκετά για να κλείσουν το κενό μεταξύ της ιδιωτικής χρηματοδότησης και της ε, δημόσιας αυτής. Έχουμε τώρα κάποιες επιτυχημένε εμπειρίες, δεν θα μπω σε πολλέ ε, λεπτομέρειες. Ε, πρέπει να ομολογήσω πως είχα ένα παράρτημα, αλλά όταν φτάσαμε εκεί στι 5-6 σελίδε, λέω ας τα αφήσουμε. Λοιπόν, έχουμε πέντε ζητήματα, πέντε τρόπους με του οποίους μπορούμε να προχωρήσουμε και μπορεί να αμυχθεί ο δημόσιο τομέα. Φοροαπαλλαγέ απλή διαδικασία, αρέσει και στις Ηνωμένε Πολιτείε και μπορούν να προχωρήσουν και να προωθήσουν την έρευνα και ανάπτυξη. Εγγυήσεις δανείων και πρωτομισιακά δάνεια και πάλι εδώ πέρα είναι, παρέχουμε χαμηλό κόστος και καλή μόχλευση αυτών των κεφαλαίων, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλα έργα υποδομών επιχορηγήσεις για να μειωθεί το αρχικό κόστος και προμήθειες, δημόσιες προμήθειες. Δεν χαρίζουμε απλά λεφτά, στοχεύουμε τα χρήματα εκεί που χρειάζεται για να αναμειχθούν περισσότερο επιχειρήσει. Ακούσαμε τη Siemens και το τι κάνουν αυτοί και το πόσο συναρπαστική τους φαίνεται η όλη διαδικασία. Μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα κονδύλια που χρησιμοποιούν αυτές οι επιχειρήσεις και τέλος, γιατί φαντάζομαι κάτι, αυτό θέλουν πολλές επιχειρήσεις να το πω και είναι μία από τις βασικές μας ε, σκέψεις για να επανέλθουμε στην, στον τομέα των αγορών και των χρήματα αγορών. Εάν δούμε τις αγορές, ένα μεγάλο βιώσιμο, ελπίζω, τμήμα της παρέμβασης για την κλιματική αλλαγή και του πρωτοκόλλου του Κιώτο, είναι η ανάγκη οι αγορές αυτές να συνεχίσουν να καθοδηγούν την ιδιωτική χρηματοδότηση σε τέτοια έργα, σε τέτοιους κλάδους. Τι θέλουν οι αγορές. Οι αγορές θέλουν εμπιστοσύνη πως θα επιζήσουν, πως θα συνεχίσουν και στο μέλλον για όλη τη διάρκεια ζωής της επένδυσης, του εξοπλισμού που χρηματοδοτούν. Αυτό έχει κρίσιμη σημασία. Οπότε ζητούν προβλεψιμότητα. Κάτι το οποίο ζητάμε συνέχεια, γιατί βεβαίω οι αγορέ άνθρακα δεν είναι πραγματικέ αγορέ, έτσι για να το πω ομά. Βασίζονται στην κρατική πολιτική. Είναι κάτι που δημιουργήθηκε για να μα καθοδηγήσει προ μια οικονομία χαμηλών εκπομπών και άρα εξαρτάται πλήρως από το πώς εξελίσσεται η οικονομία αυτή και ελπίζω, ελπίζω να έχουμε κατάληξη στην Κοπενχάγη αν και δεν το βλέπω έχουμε πολύ δρόμο ακόμα χρειαζόμαστε την πεποίθηση πως θα έχουμε κάποια κατάληξη πως θα αποτελέσουν μέλος, μέρος της λύσης οι αγορές άνθρακα επίσης ο μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης και η κοινή εφαρμογή πρέπει να απλοποιηθούν. Έχουν γίνει γραφειοκρατικός εφιάλτης. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να έχουμε δηλαδή περισσότερα έργα και περισσότερες επιχειρήσεις που θα εμπλακούν. Και η κοινή εφαρμογή και αυτή η καθαρή ανάπτυξη που ανέφερα δεν επαρκούν για το μέλλον. Πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα, χρειαζόμαστε παραπέρα βήματα. Οπότε έχουμε ίσως και πολλές πληροφορίες σε αυτή τη διαφάνεια για τους νέους μηχανισμούς. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέους μηχανισμούς με περιβαλλοντική ακαιρεότητα εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά θα γίνουν πλούσιοι αυτό πρέπει να είναι πέρα από τη νέα διαδικασία. Χρειαζόμαστε μια ακαιρεότητα. Όπως σας είπα, περιβαλλοντική πρέπει να διασφαλίσουμε πως ε, όλα τα κράτη και όλοι οι κλάδοι θα ωφεληθούν εξίσου οπωσδήποτε από ευρωπαϊκή σκοπιά ανησυχούμε για το πώς αναπτύσσονται οι μηχανισμοί, οι διαδικασίες, βλέπουμε πίεση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και όχι στους ανταγωνιστές μας. Αλλά τα ξέρετε αυτά τα έχετε συζητήσει το τελευταίο μισή έτος. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σωστές διαδικασίες συμμόρφωσης που θα είναι μετρήσιμες όσον αφορά τα αποτελέσματα. Αν λοιπόν το πετύχουμε αυτό, το τελικό μήνυμα είναι πως θα δούμε το εξής αν επιτύχουμε τους μηχανισμούς σωστά στη ζήτηση και την αγορά, την ε, αγορά άνθρακα, θα δούμε πόσο ο ιδιωτικός τομέας θα επενδύσει μόλις οι κυβερνήσεις δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο. Αλλά πρέπει να τονίσω, όπως είπαν και κάποιοι ομιλητές μας, πως πολλές από τις επενδύσεις και τις συναλλαγές που θα επηρεάσουν την κλιματική αλλαγή θα συνεχίσουν να συμβαίνουν εκτός των αγορών αυτών θα επηρεάζονται από τις κανονικές αγορές, από τις κανονικές ξένες επενδύσεις, από επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν σε νέες αγορές, χωρίς να χρειάζονται την τιμή του άνθρακα ως κίνητρο. Θα μείνω σε αυτά λοιπόν. Δεν ξέρω, ελπίζω να παρακίνησα κάποιους να διαφωνήσουν μαζί μου, να ξεκινήσει κάποια συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε χρόνο μέχρι τις 5. Σας παρακαλώ λοιπόν. Πήραμε πολλές πληροφορίες. Καλό σας ήταν που δώσαμε τη δυνατότητα στους εμπειρογνώμονες να μιλήσουν αναλυτικά. Σας παρακαλώ εσάς τώρα να είστε πολύ σύντομοι σε ερωτήσεις. Ένα λεπτό και μετά θα προσπαθήσω να σας διακόψω. Να σας καταδείξω ότι έχει τελειώσει το λεπτό. Λοιπόν, πρώτος, Κύριε Ρίπνερ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες ε, που μας έδωσαν τόσο άναπτη αναλυτικές πληροφορίες. Και οι πιο μεγάλοι σκεπτικιστές δεν πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κλιματολογική αλλαγή. Ξέρουμε ότι πρέπει να εργαστούμε υπέρ της αηφόρου ανάπτυξης. Θα πρέπει να καθορίσουμε τις προτεραιότητες, να ε, εξοικονομήσουμε τις, ε, ε, τους πόρους. Και στην ενέργεια το ίδιο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις καλύτερες δυνατές τεχνολογίες. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνετοί για να μην σφάλουμε. Είχαμε ε, στο παρελθόν φορολογικούς παραδείσους. Τώρα μπορούμε να έχουμε ίσως βιομηχανικούς παραδείσους. Πρέπει να αλλάξει ε, η νοοτροπία των πολιτών. Θα πρέπει να καταδείξουμε στους πολίτες μας ότι θα πρέπει να υπομιστούν συμπληρωματικό κόστος. Ο πλανήτης μας είναι στη διάθεσή μας μόνο για λίγο χρόνο. Η επόμενη γενιά θα τον κληρονομήσει από εμάς και θα πρέπει να τη τον δώσουμε στην ίδια κατάσταση όπως έχει σήμερα. Ερώτηση λοιπόν. Πόσα χρήματα χρησιμοποιούμε για ε, εκπαίδευση και επιμόρφωση για το θέμα αυτό. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Γκίρεκ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω προς τον κύριο Πούς Κούμαρ. Τα κοράλια στα οποία αναφέρθηκε. Εγώ δεν είμαι πεπισμένος ότι καταστρέφονται από τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί γίνεται αυτό, μήπως τα, τα νερά είναι πολύ ζεστά ή είναι πολύ όξινα. Έχουμε ένα πρόβλημα με το οποίο τα αέρια που διαλύονται στο είδο, οδηγούν στον θάνατο των οργανισμών. Δεύτερον, τα δάση απορροφούν διοξείδιο άνθρακα. και οι χημικές αντιδράσεις, χημικές αντιδράσεις επιταχύνονται. Στη Σιβηρία, παραδείγματο χάρη, βλέπουμε ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Εκεί υπάρχουν τώρα 30% περισσότερα δάση από ό,τι στο παρελθόν. Η επίδραση αυτού του νέου φαινομένου δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί. Ίσως να αυτοθεραπεύεται ε, η βιοσφαίρα. Ευχαριστώ κύριο Σπίπερ. Ναι. Νομίζω ότι περισσότεροι εμπειρογνώμονε ήταν επεπισμένοι για αυτό που έλεγαν. Παρ' όλα αυτά, έχω κάποιε ερωτήσει. Μπορείτε να μα πείτε ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής του ανθρώπου στην ε, θέρμανση του πλανήτη. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε. Δεύτερον, εδώ και 10 χρόνια δεν μειώνονται οι θερμοκρασίες ε, ε, στη γη και υπάρχουν διακεκριμένοι πυρογνώμονες που λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα μειωθούν λόγω της μειωμένης ε, ηλιακής επίδρασης, θα μειωθούν οι θερμοκρασίες. Και μετά δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί ο κύριος Στερ να αναφέρεται στις ερευνητικές επιπτώσεις των κλιματολογικών αλλαγών για τον 22ο αιώνα. Αυτό γιατί. Μετά ανησυχώ για κάτι που ελέγχθη για την ασφάλεια προγραμματισμού της βιομηχανίας. Αναλύσατε ποτέ τι θα κοστίσει αν βιαστούμε υπερβολικά. Ένα παράδειγμα στη Γερμανία. Ε, καταστράφηκαν 4 εκτάρια δάσους και εγκαταστήθηκαν εκεί μονάδες φωτοβολταϊκής ενέργειας. Ε, αυτό πόσο στοιχίζει όμως. Μετά το ΙΤΕΣ. Εάν η Ευρώπη μονομερός προχωρήσει μετά το 2013 με τις δημοπρατήσεις. Αυτό πόσο θα κοστίσει όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Το αναλύσατε αυτό στην κοστολογησή σας. Μπορώ να υποβάλω και καμιά εικοσαριά άλλες ερωτήσεις. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ μονομερής η συζήτηση και λυπούμε που δεν ακούσαμε και την άλλη πλευρά. Ευχαριστώ κύριε Καβάλιο. Thank you, uh, and Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις ε, εμπεριστατωμένες τους εισηγήσεις. Από τα όσα άκουσα, προκύπτει πως υπάρχει μια συμφωνία ότι απαιτείται χρηματοδότηση για να χρηματοδοτηθεί η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Το θέμα είναι πώς θα μοιραστούν οι συμβολές ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, καθώς και ε, γεωγραφική κατανομή του κόστους ανάμεσα στις βιομηχανοποιημένες χώρες και τις αναδυόμενες ε, ε, οικονομίες. Το επόμενο θέμα είναι πού βασικά θα πρέπει να εφαρμοστεί, μάλλον πού θα πρέπει να δοθούν τα κονδύλια. Και κάτι το οποίο είπε ο κύριος Κάμπελ είναι ότι η οικοδόμηση δυνατοτήτων είναι ε, μια επιτακτική ανάγκη στις αναπτυσσόμενες χώρες γιατί διαφορετικά ε, δεν θα έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης των χρημάτων ε, δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτά σωστά για την καταπολέμηση των κλιματικών λογών και στις βιομηχανοποιημένες χώρες ένα, μια από τις προτεραιότητες θα πρέπει να είναι η δυνατότητα, η οικοδόμηση δυνατοτήτων για την ανάπτυξη Ε, προγραμμάτων για τις, για τις ε, προηγμένες όπως είπα χώρα. Τώρα όσον αφορά την ανάπτυξη και την επίδειξη, εσείς είπατε και το αναφέρατε και στις διαφάνειές σας ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κριτήρια ουδέτερα της τεχνολογίας. Πόσο θα πρέπει να ισχύσει αυτή η ουδετερότητα. Είναι μόνο θέμα για τους παραγωγούς, για το οποίο συμφωνώ, αλλά αυτή η ουδετερότητα θα πρέπει να προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να μην γίνεται διάκριση ανάμεσα στην αιωλική, την ηλιακή και την ε, βιομάζα, να αφήσουμε τα υπόλοιπα στην αγορά. Έχουμε τα ίδια κριτήρια που θα πρέπει να ισχύσουν όταν ε, ε, μιλάμε για κονδύλια για την έρευνα και την επίδειξη. Merci, Ευχαριστώ κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές. Εγώ θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση για την Ευρώπη όσον αφορά την Ευρώπη. Στο επίπεδο της Ευρώπης έχουμε ορισμένες χώρες, κυρίως τις ε, πρώην χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ε, που έχουν ε, πολύ σημαντικές συμβολές αερίων του θερμοκηπίου όσον αφορά την ενέργεια, όπως κυρίως η Πολωνία, με εκείνες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες με βάση τον άνθρακα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στην Ευρώπη ώστε οι χώρες αυτές να περιορίσουν περισσότερο τις εκπομπές τους σε αέρια θερμοκηπίου. Δεύτερη παρατήρηση, μεγάλες υποδομές. Πώς μπορεί να βοηθήσει η Ευρώπη στους τομείς που συμβάλλουν πολύ στις εκπομπές διοξιδίου ε, αερίων του θερμοκηπίου και σκέφτομαι τον οικοδομικό κατασκευαστικό τομέα που στη Γαλλία αντιπροσωπεύει το 40% των αερίων αυτών. Πώς η Ευρώπη μπορεί να παίξει ρόλο μοχλού για την ανανέωση των ε, κτηρίων γιατί από ε, σε ορισμένε χώρε είμαστε κάπω εκεί στριμωγμένοι, α πούμε, στι κοινωνικέ κατοικίε εκεί, επίση στι συνδρομικέ εγκαταστάσει, υποδομέ. Πώ μπορούμε λοιπόν να συμβάλλει περισσότερο η Ευρώπη για τον περιορισμό των αερίων το θερμοκήπιο. Και δεύτερον, για το φόρο του άνθρακα. Ε, σε ορισμένε χώρε ε, αποφασίστηκε να, γίνει, να δημιουργηθεί αυτή η φορολογία για τα ορυκτά καύσιμα. Θα έπρεπε να μπει και η ηλεκτρισμό, κατά την άποψή μου. Αλλά ποιο απολογισμός έχει γίνει ώστε να μπορέσει ενδεχομένως να το, κάνει, να το κάνουν και άλλες χώρες. Ευχαριστώ η κυρία Χάση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας. Έχω μια ερώτηση για το θέμα των κοραλιογενών ε, υφάλων. Νομίζω πως αυτά αυτά τα πορίσματα που δείχνουν ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη για τα, τους καρολογενείς υφάλους και μια αποερήμωση των ωκεανών, πράγμα το οποίο οφείλεται στην αύξηση της θερμοκρασίας, είναι ένα από, τις, μια από τις πιο, ένα από τα πιο ανησυχητικά πορίσματα που εγώ γνωρίζω. Έχω επίσης συμμετέχει σε ακροάσιο που οι εμπειρογνώμονες έχουν πει ότι για τα κοράλια ήδη έχουμε υπερβεί το maximum όριο. ότι η μακροπρόθεσμη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα ε, στην ατμόσφαιρα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 250 ppm. Εγώ θέλω να ακούσω σχόλια για αυτό το σημείο, ιδιαίτερα από την κυρία Μαγκλέιντ και ίσως και από τον κύριο Κάμπελ αν ε, στην επιχειρηματική κοινότητα γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση για πιο φιλόδοξες, φιλόδοξους στόχους από το δύο, τους δύο βαθμούς για τους οποίους μιλάμε τώρα. Και μια ακόμα ερώτηση για τον κύριο Κάμπελ. Εσείς για τη χρηματοδότηση εστιάσατε την προσοχή σας στη δημόσια χρηματοδότηση. Όμως ε, θα ήθελα να ε, ακούσω σχόλια για άλλου είδους χρηματοδοτικές πηγές όπως φόρος ε, εκπομπών για τις διεθνείς ε, αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές. Ο κύριος Όντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσες ε, εισηγήσεις ακούσαμε και μας δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε, στο, στο, κατόφλι μιας, ενός συνόλου αποφάσεων που θα πρέπει να λάβουμε σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό επίπεδο. Θα χρειαστούν χρόνια, μα δούμε τι συμβαίνει ε, σε άλλες διαπραγματεύσεις ε, για να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία. Το βλέπουμε ήδη και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τη βιομηχανία μας, ιδιαίτερα σε έναν παγκόσμιο ιστό που ιδιαίτερα περίπλοκος γίνεται καθημερινά και μέσα από τις μεγάλες προκλήσεις αυτές που έχουμε να αντιμετωπίσουν, τι πιστεύουν οι υπηρεγνώμονές μας ε, για την ιδέα να έχουμε στα σύνορα της Ένωσης την απειλή ενός φόρου διοξιδίου του άνθρακα που θα επέτρεπε να απειλήσουμε τις άλλες περιοχές του κόσμου, εν πάση περιπτώσει να προστατεύσουμε την εσωτερική μας αγορά στις μεγάλες ε, διεθνείς διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν. Σας ευχαριστώ. Μια ακόμη ερώτηση. Από εμένα, κύριε Κάμπελ, μιλήσατε για το ότι θα πρέπει να οργανωθεί διαφορετικά το σύστημα. Ε, εννοείται δηλαδή περισσότερες δυνατότητες τι ακριβώς εννοείται. Τελευταία ερώτηση ήταν αυτή. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους ομιλητές μας. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Στέρν. Όχι βεβαίως. Αστειεύομαι. Οπότε η κυρία Μαγκλέιτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να απαντήσω μια ερώτηση που ίσως θα απαντούσε και κίνηση γρήγορα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια εκτίμηση για την εκπαίδευση και ακούγεται αυτό. Συνεχώ γνωρίζουμε πως είναι πολύ αποτελεσματική και βεβαίως εγώ θα έλεγα πως ε, ακριβώς η εκπαίδευση στη μικρή ηλικία θα έχει αποτελέσματα ως επένδυση, αλλά δεν έχω απάντηση γι' αυτό. Τώρα ας περάσουμε στα πράγματα στα οποία ε, μπορώ να απαντήσω. Η συζήτηση τώρα βεβαίω για τους κοραλιογενεί υφάλους ε, δεν είναι ακριβώ το θέμα της επιτροπή σα, Είναι η οξύνηση πράγματι των ωκεανών ο λόγος ε, για τον οποίο δεν λειτουργούν. Ε, παλαιότερα ήταν η θερμοκρασία, αλλά βλέπουμε πως ανέκαμπταν από την αύξηση της θερμοκρασίας οι ύφαλοι. Και ευχαριστώ να κάνω τη συζήτηση αυτή μαζί σας για το ότι έχουμε περάσει τώρα στη χημεία και όχι στην θερμοκρασία. Ε, πράγματι έχει σχέση ο νόμος του Χένρι, αλλά δεν είναι το μόνο το οποίο αναφέρεται. Ευχαρίστω λοιπόν να γίνει αυτή η συζήτηση. Αναφέρατε όμως γενικότερα το ζήτημα του άνθρακα στα δάση και τα φυτά και γνωρίζουμε πως ε, το να περάσουμε από τα φυτά C3 στα C4 σημαίνει πως ε, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία γίνεται λιγότερο αποτελεσματική η βιοπικιλότητα στην παχύτευση του άνθρακα. Στα επίγεια στήματα έχουμε μείωση 5%, στους ωκεανούς ε, ένα 16% ε, μείωση ε, στην αποτελεσματικότητα παχύτευση του άνθρακα. Αυτά πιο, πιο τεχνικές απαντήσεις, αλλά ευχαρίστω να επανέλθω να περάσω τώρα στην χρηματοδότηση ήλπιζα, όπως και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, βεβαίως πάντα μπορούμε να συζητάμε τις λεπτομέρειες για το ποια στοιχεία μπορούν να μειωθούν από τους παγκόσμιους μέσους όρους με διάφορες διαδικασίες, είτε μιλάμε για θέρμανση από διάφορα αέρια, είτε μιλάμε για ελαφρά ψύχρανση. Αλλά σταδιακά αυξάνεται η θερμοκρασία, δεν εξηγείται από τον ήλιο η διαφορά μεταξύ πόλων και η σημερινού, οπότε το μοντέλο αυτό ε, έχει δοκιμαστεί και έχει παραμεριστεί. Οπότε δεν έχουμε άλλη εξήγηση πλην των αερίων του θερμοκηπίου και συνεχώς ε, ε βεβαίως αυτά αυξάνονται χάρη στην ανθρώπινη παρέμβαση. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Αλλά βεβαίως ευχαριστώ να γίνει αυτή η συζήτηση μαζί σας. Ο Νίκολα Στέρν δεν είπε πως είχαμε αρνητικό αντίκτυπο, θα έχουμε αρνητικό αντίκτυπο μόνο στον 22ο αιώνα είπε πως είναι ένα μέλλον που δεν θα θέλαμε είτε μιλάμε για 6-7 βαθμούς και πως ε, δεν πρέπει να διαβούμε αυτό το κατόφλι. Και η συζήτηση είναι για τις σημερινές συνθήκες, για να μην φτάσουμε να συζητάμε για τον 22ο ε, αιώνα. Τώρα κάποιες πιο γενικές ε, απαντήσεις. Γενικά αυτό το οποίο δεν είχα χρόνο να αναφέρω είναι οι νέε συνεργίες, ε, συνεργασίες εναντί αυτού του οποίου θέλουν οι ευρωπαϊκέ εταιρείε, δηλαδή μια πιο σταθερή πολιτική όσον αφορά τον άνθρακα και, και το πακέτο αυτό ενέργεια. Και έχω πολλέ συζητήσεις τώρα με επιχειρηματίε που αισθάνονται πιο σίγουροι πώ, ακόμα και αν δεν ορίσουμε τιμή του άνθρακα ε, βλέπουν ένα μέλλον όπου θα υπάρχουν αυτές οι συνεργασίες. Το Desert Tech είναι πολύ καλό παράδειγμα. 14 συνεργασίες, 400 δισεκατομμύρια σε επενδύσεις για να έρθει η ηλιακή ενέργεια από την Βόρεια Αφρική μέσω ενός καλωδίου υψηλή τάσης στην Ευρώπη. Και αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα. Αυτές οι συνεργασίες δεν θα τις είχαμε σκεφτεί καν πριν από ένα-δύο χρόνια. Έχουμε τώρα κατασκευαστές αυτοκινήτων, ε, οχημάτων που συζητάνε στην Δανία την δυνατότητα ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, ε, συνεργασίες που δεν θα υπήρχαν. Οπότε συνεργασίες ε, δημόσιο ιδιωτικού τομέα, δηλαδή δημόσια αγαθά με το κίνητρο του κέρδους λίγο παρακάτω. Ακούω βεβαίως μια ελευθερία απογοήτευση για το ότι οι νέοι αυτοί τρόποι επενδύσεων απαιτούν αυτή τη σταθερότητα μπορεί να δώσει μόνο η δημόσια επένδυση. Οπότε, ε, για να επανέλθω στο στο σχόλιο που έκανα για τα πακέτα δημοσιονομικής διάδοσης. Είναι φοβερά τα ποσά που ξοδεύονται στην ανακαίνιση κτηρίων. Στην Αυστρία, π.χ. για την θερμική ανακαίνιση κτηρίων, δημοσίων κτηρίων, 345 εκατομμύρια. Τσεχία, 900 εκατομμύρια. Γαλλία, 200 και τα λοιπά και τα λοιπά. 3 ε, δισεκατομμύρια στη Γερμανία για τη βελτίωση των δημοσίων κτηρίων και μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών. Οπότε υπάρχει στόχευση στα κτίρια, αλλά όχι συγκεκριμένα στην ανακαίνιση. Πάνε στα εύκολα πράγματα που μας δίνουν ε, γρήγορο κέρδος. Εκεί που δεν ε, θεωρεί η βιομηχανία ότι θα υποφεληθεί είναι το φαινόμενο ανάκαμψης που θα υπήρχε. Δηλαδή αν γίνονταν πιο Αποτελεσματικέ στην ενέργεια, η εξοικονόμηση αυτή δεν μένει εντό τη εταιρεία. δεν υποφελείται η εταιρεία. Οπότε βλέπουμε τώρα μεγαλύτερη ζήτηση για έρευνα και ανάπτυξη για να υπάρχουν αυτέ οι συνεργασίε, για να υπάρξει επένδυση στον χαμηλό ανθρακά. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Η ισορροπία λοιπόν μεταξύ των νέων αυτών πακέτων και του να δώσουμε κίνητρα στην καινοτομία. Τώρα, αν πιστεύω σε φόρο άνθρακα, είναι πολύ σημαντικό μήνυμα προς τους καταναλωτές, γιατί οι καταναλωτές αυτή τη στιγμή δεν αισθάνονται την πίεση στο σημείο, στη στιγμή της αγοράς. Εκεί πέρα μας λείπει κάτι. Βεβαίω το εύκολο για να γίνει είναι ε, στα ανάντι που λέμε, στον παραγωγό της ενέργειας. Οπότε πρέπει να δούμε το τι κάνουμε και παγκόσμια και ως Ευρωπαίοι αλλά και τη στιγμή τη αγορά για να αντιληφθούν τη σύνδεση ανάμεσα στου πόρου τον άνθρακα και το πόσα λεφτά έχουν ή δεν έχουν στην τσέπη του οι καταναλωτές. Οπότε νομίζω η Επιτροπή Στέρν έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά για να ξεκινήσει το πώς μεταφράζεται αυτό στι τσέπε των ανθρώπων αλλά πρέπει και τα και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί να ετοιμαστούν για να δώσουμε κίνητρα προς τα ανάντη και φορολογία προς τα κάτω. Επίσης υπήρχε μια πάρα πολύ καλή μελέτη για το πώς ωφελούμαστε με το να πετύχουμε σωστά τα πράγματα. Αν όμως προσθέσουμε όλα τα περιβαλλοντικά μειονεκτήματα των ε, ορικτών καυσίμων έχουμε 6 ευρώ ανά κιλοβατόρα ενώ οι ανανεώσιμες πηγές είναι 0,8 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Οπότε με αυτά τα νούμερα θα σας αφήσω, γιατί και πάλι χρησιμοποιούνται από την ίδια τη βιομηχανία για να αλλάξουν την εσωτερική του αγορά, για το πώς θα χρεώνουν ο ένας τον άλλον. Και βεβαίως και στα προϊόντα τα οποία παρέχουν στο κοινό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Σκέμπελ έχει το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους βουλευτές για τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσει που μου υπέβαλαν. Μερικέ από αυτές θα χρειαζόμουν μια εβδομάδα για να σας απαντήσω. Θα προσπαθώ να αναφερθώ στις άμεσες προς την και κάποια σχόλια που ζητήθηκε μου συζητήσατε να σχολιάσουμε ποια ποσοστά είναι υπεύθυνα για τις κλιματολογικέ αλλαγές. Αν διαβάσετε τη βιβλιογραφία θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά μέτρα που παίζουν ένα ρόλο και κατά βάση είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι αναπτυσσόμενες χώρες. είναι εκείνες που θα πρέπει να αναλάβουν τον ηγετικό ρόλο για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τα προβλήματα. Και οπωσδήποτε από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αναλάβει την ηγεσία. Και η ανησυχία μου είναι να κοιτάξουμε πίσω μα να δούμε ποιο μα ακολουθεί έχουμε ξεκινήσει, αλλά θα πρέπει να έρθουν πιο κοντά σε εμά. Και περνάω εδώ σε μια ερώτηση που υπευλήθη όσον αφορά την αναγουστικότητα και το θέμα του φόρου στα σύνορα. Η επιχειρησιακή Ευρώπη είναι βέβαια υπέρ των ανοιχτών αγορών, ορισμένα τα μέλη μας, οι Γάλλοι ιδιαίτερα, ανησυχούν και θεωρούν ότι ίσως η απειλή των συνοριακών φόρων θα, έχουν, θα έχει επιπτώσεις στις διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρω αυτό είναι αληθές ή όχι. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι θα, ε, θα προωθήσει τις ε, εισαγωγές. Θα είναι πολύ δύσκολο νομίζω να καταμετρήσουμε τις επιπτώσεις οι δύο βιομηχανίες που επιμένουν, τσιμέντο και αχάλιβα, ίσως θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, δεν ξέρω, θα πρέπει να το δούμε αυτό. Γίνονται πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό στις ε, διαπραγματεύσεις. Η κυρία Χάση αναφέρθηκε στο θέμα των ε, ε, φόρων για τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό είναι πάλι ένα θέμα ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, γιατί φοβούνται ότι άλλοι φορείς θα εκμεταλλευτούν το θέμα. Παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις. Εγώ ήμουν στην Βαρκελόνη προσεκτικά και είδα να υπάρχουν διαφορετικές ε, κινήσεις κατά πόσον οι κλιματολογικές αλλαγές ε, αφορούνται από τις μεταφορές ε, της Νενέρης και της ε, θαλάσσιας. Δεν ξέρω τελικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά μπορώ να σας α, διαβεβαιώσω ότι πραγματικά είχε σκληρύνει το παιχνίδι όταν γινόντουσαν οι διαπραγματεύσει αυτέ. Και είναι θέμα στο οποίο θα μπορούμε να επανέλθουμε βέβαια. Έχει όμω πάρα πολύ έντονο ανταγωνιστικό ενδιαφέρον για τι ε, ευρωπαϊκέ αεροπορικέ εταιρείε. Η κυρία Καβάλο υπέβαλε μια σειρά ερωτήσεων. Η μία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν ήταν ερώτηση, αλλά ανάφερε στην δημιουργία δυναμικού. Ένα από τα κύρια θέματα στο οποίο νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στον τομέα κλιματολογικών αλλαγών στην Κοπενχάγη είναι τα τεχνολογικά συμβουλευτικά κέντρα. Εκεί μπορεί να υπάρχει δημιουργία δυναμικού, αλλά είναι επίσης μια πρόορη κίνηση για την ανάπτυξη των κέντρων αυτών και αν παρακολουθήσει κανένα εξελίξει, παραδείγματο χάρη χρήση τη ενέργεια, σκεφτείτε πόσε οικονομίε μπορούν να γίνουν αν έχουν τοποθετηθεί περιφερειακά για να λαμβάνουν υπόψη οι περιφερειακές διαφορές και συγκεντρώστε την προσοχή σε ένα θέμα, όπως είπε και η κυρία Μακρέιτ, μπορεί να υπάρχει μεγάλη επιτυχία, μεγάλες αλλαγές, παραδείγματος χάρη η ανακαίνιση κτίριων στην Ευρώπη, η αναγέννηση κτίριων αλλού στον κόσμο. Κάτι τέτοιο θα κόστησε λίγα χρήματα, Ευρωπαϊκή Ένωση το υποστηρίζει, οι Ηνωμένε Πολιτείε το υποστηρίζουν, η Ιαπωνία ξεκίνησε. Εκεί λοιπόν υπάρχει έντονη στήριξη και μπορούμε να προχωρήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα τη δική σας ερώτηση. Ίσως θα πρέπει να την ξαναυποβάλλετε. Κατά τα άλλα, κάλυψα όλε τι αποπτώσει. Α, όχι, το τελευταίο σημείο, κατά πόσο πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ των τεχνολογιών. Πάλι, ισορροπία θα υπάρχει. Το μόνο που θα πετύχουμε θα είναι μια ισορροπία. Υπάρχουν πλεονεκτήματα για οτιδήποτε. Ε, λοιπόν, η εστίαση στις βιομηχανίες να γίνει χωρίς να αντιτελεχθεί όμως η ισορροπία που έχει επιτευχθεί. Παραδείγματος χάρη ε, ξεκινά το θέμα της, σε μια άλλη αίθουσα, εδώ συζητιέται το θέμα της ε, εξουδετέρωσης των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από την ηλεκτρική τη βιομηχανία παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια κλιματολογικών ενεργών και θα σταματήσω, Πρόεδρε. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σκόμα, νομίζω ότι δόθηκαν οι περισσότερε απαντήσει από του άλλου εμπειρογνώμονε. Αλλά υπάρχουν δύο πράγματα που εγώ θα ήθελα να αναφέρω εδώ. Ε, αναφέρθηκε το ερώτημα από τον κύριο Μπίρμπεργκ για το ποιο ποσοστό των κλιματικών αλλαγών μπορεί να αποδοθεί στους ε, ανθρώπους ή στις ε, ανθρώπινες δραστηριότητες. Αν δούμε τα φαινόμενα, να δούμε την μεγάλη κλίμακα των τελευταίων 20.000 χρονών, θα βλέπαμε ότι είναι ασφαλές να συμπεράνουμε πως οφείλονται στην ανθρώπινη παρέμβαση και δραστηριότητα. Ακόμα και αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πάντως λέω πως είναι, είναι σίγουρο το να το πούμε για διάφο, πολλούς και διάφορους λόγους. Κάτι άλλο που ρωτήσατε αφορά τα κοράλια Όμως ε, κάτι που αφορά τους κοραλιογενείς υφάλους που είναι νέο εξάλλου στοιχείο για την ομάδα μας στην Καραϊβική θάλασσα, στην Ειρηνικό κενό είδαμε ότι ε, ε, περισσότερες δραστηριότητες εκεί είναι αλληλεία χωρίς ε, ιδιαίτερη προστασία, παράκτια προστασία και τουρισμός που προσθέτουν, ε, επιβαρύνουν τις περιοχές αυτές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν κάποιες δράσεις για να προστατευτούν τα κοράλια, όχι προς χάρη μόνο των πράσινων ε, ανησυχιών, αλλά και για να απομακρυνθεί η φτώχεια από αυτές τις περιοχές. Δεν έχω σημειώσει κάποια άλλη ερώτηση την οποία απευθύνεται σε μένα. Η μετακίνηση των κλιματικών αλλαγών ε, ε, ε, αναφέρθηκε για τη μετακίνηση του φόρτου, του βάρους το κακό που εμείς κάνουμε και το μεταφέρουμε στις μελλοντικέ γενναίες. Αυτό ήταν το πλαίσιο βασικά. Η Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βουδηματά, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, για τις πληροφορίες. Δεν θέλω να πω την τελευταία φορά που θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Μετά από μια σύντομη διακοπή θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Εντάξει. Ναι. Σας ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισε. να μην σας ξαναχαιρετήσω βέβαια. Το επόμενο σημείο τη εμερησίας διάταξη είναι το 11. για τη χρήση βιοκτώνων προϊόντων. Έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων προβλέψει σήμερα. Ο εισηγητή είναι ο κύριος Καρίμ, ο οποίος είναι εδώ. Και θα σας ήμουν ευγνώμων να αρχίσετε κύριε Καρίμ. Όλοι όσοι οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν στην αίθουσα, αλλά κάτι έχουν να συζητήσουν, παρακαλώ να βγουν από την αίθουσα. Can start with our work. Thanks. Um, Πρόεδρε, συνάδελφοι, εγώ θα μιλήσω για αυτό το θέμα της εμπορίας βιοκτώνων. Σήμερα είναι βεβαίως η ανταλλαγή απόψεων επί του θέματο. Οι άλλες σημαντικές ημερομηνίε που θα πρέπει να σημειώσουν οι συνάδελφοι είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 26 Ιανουαρίου του επόμενου έτος Και η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 22-23 Φεβρουαρίου με ενδεχόμενη ψηφοφορία στην Ολομέλεια, ελπίζω, τον Μάιο το επόμενου έτος. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Τώρα, σε σχέση με το θέμα αυτό, θα πρέπει να σας πω ότι όταν, να σας ομολογήσω ότι όταν ανέλαβα το συγκεκριμένο θέμα δεν ε, είχα εκτεταμένη γνώση των βιοκτώνων προϊόντων ή ε, το πώς ακριβώς λειτουργούν και είμαι βέβαιος το ίδιο θα συμβαίνει και με πολλούς συναδέλφους. Ε, όμως, από ό,τι κατάλαβα εγώ και το έχω μελετήσει, η συντομία είναι η εξή. Είμαι νέο μέλο αυτή εδώ τη Επιτροπή, αλλά υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν συνεργαστεί μαζί μου παλιότερα και θα γνωρίζουν ότι όταν είχα να συντάξω εκθέσει ή γνωμοδοτήσει σε άλλε επιτροπέ, εγώ κρατούσα πάντοτε τι πόρτε ανοιχτέ. Είμαι δηλαδή ανοιχτό στο να ακούσω τι απόψει των συναδέλφων, να τι συζητήσω για να δούμε πώ θα προχωρήσουμε. Τα βιοκτώνα προϊόντα είναι ενεργές ουσίες όπως χημικές ουσίες ή μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν οργανισμούς που είναι βλαβεροί όπως για παράδειγμα είτε για την ανθρώπινη υγεία είτε για την ζωική υγεία. Χρησιμοποιούνται για να προστατέψουν προϊόντα από οργανισμούς που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά. Και παραδείγματα είναι τα απολυμαντικά μέχρι τα προϊόντα που ελέγχουν την, τους, τα, έντομα. Έχουμε την οδηγία για τα βιοκτώνα που εισήχθη πριν κάποιο καιρό με διπλό στόχο καταρχήν την εισήγηση, την, ε, μάλλον την προστασία του περιβάλλοντος και δεύτερον τη δημιουργία ενός ε, πλαισίου, μιας δομής μέσω της οποίας οι νέες ενεργές ουσίες και προϊόντα θα εγκρίνονταν. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα, η οδηγία πιστεύω δεν ήταν ε, αποτελεσματική καθόλου υπήρξε μόνο μία νέα ενεργεία ουσία, η οποία μόλις εγκρίθηκε με βάση το ισχυόν σύστημα και μόνο 30 ουσίες εν γέννη, συνολικά μάλλον, ε, υπάρχουν στον κατάλογο της Ένωσης για τα επιτρεπόμενα προϊόντα. Πρότασή μου είναι να ευθυγραμμιστεί η ισχύουσα διαδικασία και να αυξηθεί η σαφήνεια των απαιτήσεων για τι ενεργέ ουσίε και για τα βιοκτώνα προϊόντα. Επίση, προσπαθώ να εισάγω περαιτέρω προστασία για το περιβάλλον. Πιστεύω πως ε, η Κομισιόν ε, κάνει κάποιες καλές προτάσεις μέσω αυτής της έκθεσης. Μια πρόταση για μια κεντροποιημένη διαδικασία αδειοδότησης που θα την αναλάβει η CEJ για τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου καθώς και ένα βελτιωμένο σύστημα αμοιβέ συνεργασία σε όλα τα κράτη-μέλη θα βελτίωναν την ε, ισχύουσα διαδικασία και θα ενθάρρυναν την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Βεβαίω, ε, Πρόεδρε, η προστασία του περιβάλλοντος ε, θα πρέπει να είναι πρώτη στη μας ε, μέρημνα, όμως θα πρέπει η νέα νομοθεσία να παρέχει ένα πλαίσιο το οποίο να είναι λειτουργικό για τον κλάδο και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να παρέχει κίνητρα για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα αυτό το, η αγορά των βιοκτώνων προϊόντων είναι πολύ μικρότερη από αυτή των, ε, των, των ζενιοκτώνων και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της δημόσιας υγείας. Υπάρχουν διαφορετική, έχουν διαφορετική χρήση από ό,τι τα ζενιοκτώνα, αν και κάποιες φορές ε, περιέχουν τα ίδια χημικά. Κάποιοι τομείς της πρότασης πιστεύω θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά κατά πόσο το εύρος του προϊόντος χαμηλού κινδύνου που θα πρέπει να το αναλάβει και μια κεντρική, ένας κεντρικός οργανισμός είναι, στο, είναι σωστός. Δεύτερον, κατά πόσο τα κριτήρια αποκλεισμού θα πρέπει να προσαρμοστούν. Τρίτον, αν ε, το κόστος της διαδικασίας της αδειοδότησης που προτείνει η Κομισιόν είναι λογικό και λειτουργικό για την ε, βιομηχανία. Και μετά έχουμε και το θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης. Και τέλος, αν το πεδίο της χρήσης επιτροπολογίας, όπως προβλέπετε από την πρόταση, είναι σωστό. Πρόεδρε, ε, πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ελπίζω να σας εξέθεσα με σαφήνεια τις αρχικές μου απόψεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα για να συντάξουμε τη γνωμοδότηση αυτή και σίγουρα θα ήθελα να καλέσω τους ε, συναδέλφους να συμβάλλουν εδώ είτε σήμερα είτε αργότερα και αυτό είναι αποδεκτό. Και από αυτή τη βάση πρόεδρε μπορείτε να ξεκινήσετε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Πατριτσέλο έχει ζητήσει το λόγο. Εγώ θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή Καρίμ για την ε, εισήγησή του. Και θέλω να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για τη δουλειά που έκανε μέχρι στιγμή στην εκπόνηση μια νομοθετική πρόταση που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και σύμμορφη με του στόχου που σκοπεύει να επιδιώξει ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία τη ανθρώπινη υγεία. Φυσικά πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο διάβασα με μεγάλη προσοχή και εκτίμησα το γενικό του χαρακτήρα αλλά φαίνεται πω ορισμένα στοιχεία ειδικά μπορεί να βελτιωθούν ιδιαίτερα με στόχο να μην επιβαρύνουμε με περιτά βάρη τις μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αυτήν, ε, ε, στο πλαίσιο το οποίο καλύπτει η οδηγία. Η οδηγία η προηγούμενη θα αντικατασταθεί από έναν κανονισμό, όπω προβλέπει η Κομισιόν. Αυτό θα επιτρέψει να υπάρχει μια ίση και άμεση εφαρμογή όλων των προδιαγραφών, όλων των διατάξεων από τα κράτη-μέλη, ενώ θα ξεπεραστεί ανάγκη να υπάρχει μια μεταβατική περίοδο και μέτρα υποδοχής που είναι απαραίτητα να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο. Ένας κανονισμός λοιπόν θα μας εγγυηθεί μια καλύτερη εναρμόνιση της ευρωπαϊκής αγοράς, θα απλοποιήσει εξάλλου τα διοικητικά κόστη για τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά την διαδικασία διοδότησης, εγώ δέχομαι με μεγάλη ικανοποίηση τη δυνατότητα να υπάρχει μια κεντρική αδειοδότηση που θα την διαχειρίζεται άμεσα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις χημικές ουσίες, για τα βιοκτώνα ε, που περιλαμβάνουν νέες ε, ενεργές ουσίες και βιοκτώνα χαμηλού κινδύνου. Είναι απαραίτητο μια τέτοια διαδικασία να επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, ακόμα και για τα βιοκτώνα υψηλού κινδύνου, εφόσον αυτό θα εγγυόταν μια καλύτερη λειτουργία τη εσωτερική αγορίας και θα διευκόλυνε του παραγωγού που λειτουργούν στι διάφορε εθνικέ αγορέ. Επιπλέον, συμμερίζομαι απόλυτα την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνοδεύσει την κεντρική διαδικασία από μια διαδικασία εθνική ε, αδειοδότηση. Αυτό αποτελεί μια, έναν επιπλέον, μια επιπλέον προστασία για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει που λειτουργούν στον τομέα αυτό και που είναι πολυάριθμες και είναι βασικά αυτές που θίγονται και από την οικονομική κρίση, γιατί έτσι δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στην εθνική διαδικασία διαδότησης και εκείνη την κεντροποιημένη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού πάντοτε με βάση για την αδειοδότηση είναι δίκαιο οι ενεργές ουσίες να αποτελέσουν αντικείμενο αυστηρής αξιολόγηση όσον αφορά τους κινδύνους για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον πριν να συμπεριληφθούν στο παράρτημα 1. Αλλά αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από μια συγκριτική αξιολόγηση, όπως προβλέπει το άρθρο 21 του κανονισμού, με δημιουργεί έτσι ένα δεύτερο επίπεδο ε, αξιολόγηση των ενεργών νησιών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και το θέμα των ε, τιμών, του κόστου, με υπό το φω των διαφορών που υπήρξαν τα παλιότερα χρόνια ανάμεσα στο κόστο αξιολόγηση τη ενεργού ουσία ε, στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρχει ένα εναρμονισμένο σύστημα κόστου τιμών που θα εμποδίζει την κερδοσκοπία, πράγμα το οποίο βλάπτει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα πρέπει να εγγυηθούμε ένα καθεστώ συναρμονισμένο και συνεπές. Όσον αφορά την ετικετοθεσία, ευνοϊκά διακύμεθα στις νέες διατάξεις που θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να προβούν σε επιλογές γνωρίζοντας ε, τα συστατικά και καταργώντας ε, τις διακρίσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους Ευρωπαίους και τους αλλοδαπούς ε, παραγωγούς. Ε, θεωρεί, θεωρώ πως είναι περιττό, τον αναφέρεται στην ετικέτα ο αριθμός αδειοδότησης όλων των βιοκτώνων. Θα ήταν αυτό μια επικάλυψη με άλλες νομοθεσίες που δεν θα αποφέρουν κανένα όφελος ούτε στο περιβάλλον ούτε στην ανθρώπινη υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Κατόπιν η συνάδελφος κυρία Ριβάζη έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια πως είναι ενδιαφέρον το πέρασμα από οδηγία σε κανονισμό. Όχι τόσο γιατί ευνοείται σε επιχειρήσεις, αλλά για να υπάρξει εναρμόνιση σε κάθε κράτος. Γιατί ανάμεσα στα κράτη που μεταγράφουν γρήγορα και τα κράτη που κάνουν χρόνια για να μεταγράψουν μια οδηγία, βλέπουμε πως αυτό δεν βοηθά και πολύ το εσωτερική αγορά. Εγώ θεωρώ πως θα πρέπει να φτάσουμε σε μια συνοχή ανάμεσα στα όσα κάναμε για τα ζυζανιοκτώνα και όσα θα κάνουμε για τα βιοκτώνα. Αυτή η συνοχή είναι πολύ σημαντική και νομίζω πως υπάρχουν δύο σημεία κλειδιά σε αυτή τη νέα νομοθεσία που θα πρέπει ίσως να τα λάβουμε υπόψη. Το πρώτο είναι η ευθύνη των κρατών μελών στην αδειοδότηση προϊόντων και το δεύτερο είναι τα κριτήρια αποκλεισμού για τις ενεργές ουσίες. Το πρώτο σημείο, ευθύνη των κρατών μελών στην αδειοδότηση των προϊόντων. Φαίνεται πως σε αυτήν την νομοθεσία υπάρχει δυνατότητα ε, μη έγκρισης από ένα κράτος μέλος. Όταν όμως πρόκειται για τα ζυζανιοκτώνα, ήταν δυνατόν ένα κράτος μέλος να αρνηθεί την έγκριση, την αδειοδότηση. Ενώ για τα βιοκτώνα κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία υποχρεωτική αμοιβαία αναγνώριση. Και από τη στιγμή που υπάρχει αμοιβαία υποχρεωτική αναγνώριση, ισχύει για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα μια χώρα να τα αρνηθεί την αδειοδότηση. Και αυτό δεν ίσχυε για τα ζενιοκτώνα. Δεύτερον, οι προϋποθέσεις για την προσαρμογή στις τοπικές περιστάσεις. Για τα ζενιοκτώνα δεν υπήρχαν όροι, δεν υπήρχαν προϋποθέσεις, ενώ για τα βιοκτώνα υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις και όροι. Άρα λοιπόν ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να τροποποιήσει μια αναδιοδότηση σε σχέση με, τις, ε, με βάση μάλλον τις τοπικές ε, περιστάσεις. Και έπειτα, στην δυνατότητα περιορισμού της χρήσης, ε, στην περίπτωση των ζενεκτών ήταν δυνατόν, στα βιοκτώνα δεν γίνεται πλέον δεν είναι πλέον δυνατόν. Ενώ ορισμένε χώρε μπορεί να έχουν ε, διαφορετικέ χρήσει ανάλογα με την ε, νοοτροπία τη κάθε χώρα. Και έπειτα για την κεντρική αδειοδότηση, για τα ζυζανιοκτώνα δεν, δεν γινόταν αυτό, ενώ τώρα ναι για τα βιοκτώνα. Φαίνεται λοιπόν ότι στην επιχειρηματολογία για τα βιοκτώνα είμαστε πολύ πιο περιοριστικοί όσον αφορά την κυριαρχία των κρατών. Και ότι έχουμε πολύ περισσότερες δυσκολίες να τροποποιήσουμε την έγκριση, να διαδότηση. Θα πρέπει λοιπόν αυτά κανονικά να ε, εναρμονιστούν. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο συνεπές. Δεύτερον, κριτήρια αποκλεισμού των ενεργών ουσιών. Δεν θα πω στις λεπτομέρειες, αλλά αν δει κανείς από ε, τις λεπτομέρειες της οδηγίας, ορισμένα κριτήρια που ίσχυαν για τα ζενοκτώνα δεν προτείνονται για τα βιοκτώνα, ενώ με, ε, είναι οι ίδιες ουσίες, με ίσως διαφορετικό βαθμό συγκέντρωσης. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι περίπου 50.000 προϊόντα υπάρχουν που περιλαμβάνουν βιοκτώνα, δηλαδή ε, μπορεί να είναι για προϊόντα υγιεινής, απολύμασης κτλ. Και τα άδαμε κάποια κινέζικα προϊόντα που ήρθαν στη Γαλλία και που δεν υπέστησαν κανέναν άλλο έλεγχο και δημιούργησαν προβλήματα όλα όσα είναι επίμονα, βιοσορευτικά, τοξικά, εξαιρετικά επίμονα ή ρηπογόνα και πολύ επίμονα ε, δεν υπάρχουν εδώ ως κριτήρια στα βιοκτώνα ενώ υπήρχαν στα ζενιοκτώνα. Αυτό θα πει μαζί με τα υπόλοιπα που σας είπα. αυτά που ήθελα να πω για τα κριτήρια αποκλεισμού βρίσκω ότι στο επίπεδο των βιοκτών είναι λιγότερο αυστηρά είναι λίγο πιο ελαστικά και δεν είναι αρκετά συγκεκριμένα, δεν είναι καλά ορισμένα. Κύριε Σιγητά, λοιπόν, θα πρέπει να δείτε, να προσέξετε ώστε να υπάρχει καλύτερη προστασία απέναντι στην υγεία, γιατί είναι προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα. Και έπειτα είχαμε πρόταση να σας κάνω, δηλαδή να ε, εισάγετε και τα νανοσωματίδια γιατί η χρήση τους είναι εξαιρετικά διευρυμένη, είναι ανεξέλεγκτη και δεν περιλαμβάνεται στην ετικετοθεσία. Ήταν μια από τις προτάσεις του εισηγητή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για αυτόν τον κανονισμό. Την πρόταση κανονισμού μάλλον. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις σύντομες και ακριβείς ε, τοποθετήσεις σας. Κατόπιν η Κομισιόν έχει το λόγο η κυρία Κουτσί, ελπίζω να είπα σωστά το όνομά σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις κυρίες και του κυρίους βουλευτές που έκαναν χρήσιμα και επικοδομητικά σχόλια. Ευχαριστώ τον κύριο Καρίν ε, για την ενδιαφέρουσα αυτή πρόταση είναι ενδιαφέρουσα γιατί υπήρχε νομοθεσία ε, εδώ και 7-8 χρόνια και θέλουμε να λειτουργήσει και ο κύριος Καρίν τόνισε τις ελλείψεις της ε, ε, κείμενης νομοθεσίας. Οπότε θέλουμε απλά να απλοποιήσουμε την διαδικασία γιατί ο κλάδος αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις οπότε αν απλοποιήσουμε και ξεκαθαρίσουμε τις προθεσμίες θα είναι κάτι πολύ σημαντικό και βέβαια ο βασικός στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος ε, και της υγείας ήδη στην οδηγία. Ξέρουμε πως υπήρχαν όμως παραθυράκια όπως η σήμανση ε, κατεργασμένων εισαγόμενων ειδών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ουσίες που δεν επιτρέπονται καν στην Ευρώπη σε αυτά τα είδη και είχαμε πολύ σοβαρές βλάβες ε, προς τους ε, καταναλωτές. Οπότε τα είδη στο μέλλον πρέπει να έχουν σαφή σήμανση. Θα εισάγονται μόνο είδη με ουσίες που επιτρέπονται στην Ευρώπη, οπότε θα προστατεύονται σωστά οι καταναλωτές. Επίσης, όπως τόνισαν κάποια μέλη, διασφαλίσαμε πως κάποια από τα προϊόντα πηγαίνουν στην κεντρική διαδικασία που βεβαίως είναι πιο αποτελεσματική και πρέπει να απλοποιήσει την άδεια και προτείναμε να μην εφαρμοστεί αυτό για όλα τα προϊόντα γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως σε αυτή την αγορά έχουμε χιλιάδες προϊόντα που έχουν λάβει άδεια στα κράτη-μέλη και το να γίνει αυτό από τη μια μέρα στην άλλη να πάει σε μια νέα υπηρεσία, σχετικά νέα, ίσως παρά είναι. Και πρέπει να λειτουργεί και το σύστημα και να ενδιαφερθούν και εταιρείε να πάνε στο, στην κεντρική αυτή διαδικασία. Γι' αυτό διαλέξαμε το εξής. Μια κεντρική διαδικασία για όλα τα προϊόντα που αποτελούνται από νέες ουσίες. Όχι αυτά λοιπόν που κυκλοφορούν τώρα, αλλά αυτά που θα αναπτυχθούν από εταιρείε αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή και μετά θα γίνουν κάποια προϊόντα και, τα, και για τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου. Βεβαίω είναι σημαντικός ο ορισμός του χαμηλού κινδύνου και μπορεί να τον ξεκαθαρίσουμε στις ε, συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Γιατί τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου, γιατί θέλαμε οι εταιρείε να ενδιαφερθούν να διαθέσουν προϊόντα στην αγορά στο μέλλον που θα, έχουν, θα αντιπροσωπεύουν χαμηλότερο κίνδυνο από τα προϊόντα που πολλούνται αυτή τη στιγμή. Βέβαια, πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην πράξη, αλλά εμείς το είδαμε ως ένα κίνητρο. Μετά για τα τέλη. Άκουσα από τον κύριο Καρίν πως πρέπει να εναρμονιστούν. Νομίζω η δομή πρέπει να εναρμονιστεί σε εθνικό επίπεδο η δομή των τελών δύσκολο θα είναι να το προτείνουμε εμείς αν δεν το περιέχει η πρόταση γιατί κάθε δημόσια αρχή έχει διαφορετικό κόστος οπότε πρέπει να αφήσουμε ελευθερία στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν το ύψος αλλά πρέπει να αναμονιστεί η δομή να υπάρχουν δηλαδή οι ίδιοι κανόνες σε όλη την Ευρώπη και βεβαίως για αυτά που τα τέλη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χημικών αυτά είναι πανευρωπαϊκά και αποφασίζονται από την Επιτροπολογία σύμφωνα με το ΡΙΤΣ. Τώρα για την συνοχή μεταξύ εντομοκτώνων και ζυζανιοκτώνων και βιοκτώνων πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο κλάδων όπως τόνισα στις άλλες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Ο τομέας των ζυζανιοκτώνων σχετίζεται αποκλειστικά με τη γεωργία και άρα με τοπικές συνθήκες. Όταν μιλάμε όμως για βιοκτώνα, όπως είπε και ο κύριος Κάριμ, μιλάμε για πολύ πολλούς διαφορετικούς βιομηχανικούς ε, τομείς που είναι από τα υφαλοχρώματα πλοίων μέχρι απολυμαντικά, εντομοκτώνα, διαφορετικά πράγματα. Και οπότε δεν δικαιολογείται να έχουμε τοπικές συνθήκες για όλους αυτούς τους ε, κλάδους. Μπορεί να υπάρχει κάποια συνοχή, αλλά όχι παντού. Από την άλλη, επειδή θέλουμε βεβαίως μια εσωτερική αγορά που θα λειτουργεί καλύτερα για να μειώσει το κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλήθεια είναι ότι έχουμε ενισχύσει την αμοιβαία αναγνώριση, ακριβώς για να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και γιατί νομίζουμε πως σε πολλές περιπτώσεις δεν ισχύουν οι τοπικές συνθήκες. Παρόλα αυτά, τα κράτη-μέλη μπορούν να γύρουν κάποια αντίρρηση στην αμοιβαία αναγνώριση αν δεν θεωρούν ασφαλές το προϊόν ή αν υπάρχουν τοπικές συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε αυτό. Και τέλος για τα κριτήρια αποκλεισμού πράγματι μας ανησυχεί το ότι οι ουσίες που λέμε πιο επικίνδυνες δεν θα επιτραπούν. Ε, πρέπει πράγματι να δούμε τη συνοχή με την νομοθεσία των ε, ζυζανιοκτώνων, με αυτό συμφωνώ. Αλλά υπάρχει πράγματι μία λογική στο να έχουμε πολύ αυστηρά κριτήρια για τα βιοκτώνα με μία εξαίρεση ίσως γιατί υπάρχουν καταστάσεις γιατί μιλάμε για κλάδους βιομηχανίας όπου για λόγους δημόσιας υγείας ή γενικούς περιβαλλοντικούς στόχους ίσως να μην είναι σωστό να χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια αποκλεισμού. Οπότε η εξαίρεση της εξαίρεσης δηλαδή θα ε, είχε εφαρμογή στα βιοκτώνα αλλά βεβαίως είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε και τέλος για τα νανοσωματίδια. Βεβαίως η αξιολόγηση κινδύνου καλύπτει τα πάντα και τα νανοσωματίδια είναι προφανές. Ακούσαμε πώ είχαμε ειδικέ διατάξεις για τα νανοσωματίδια. Εμεί θεωρούμε πως δεν είναι αναγκαίες ειδικά για τα νανοσωματίδια γιατί η αξιολόγηση κινδύνου καλύπτει και τον κίνδυνο και την έκθεση και την φύση της ουσίας αλλά βεβαίως μπορούμε να το δούμε. Αυτά ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα επικοδομητικά σας σχόλια και αναμένουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο και ο συζητής και ο έχει συζητήσει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, εγώ Συμφωνώ με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι που προηγήθηκαν και με τον εισηγητή για τα όσα λέει αυτή η πρόταση κανονισμού. Εγώ πιστεύω πως ε, Μια μεγαλύτερη σύνεση δεν ε, θα βλάψει κανέναν. Εγώ τα είδα όλα αυτά με πολύ προσοχή και πιστεύω πως πολλά θέματα που εκ πρώτης απόψεως μπορεί να προκαλούν ε, ανησυχία ξεπεράστηκαν και από το... τα όσα μας είπε εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ακούσαμε κάποια πράγματα για τα οποία χρειάζεται διευκρίνηση. Χρειαζόταν μάλλον διευκρίνηση. Δύο σύντομες ερωτήσεις θέλω εγώ να θέσω για να μπορέσουμε καλύτερα να αξιολογήσουμε το θέμα. Στο άρθρο 47, όταν μιλάμε για την εμπορία ή για το προϊόν ή για το υλικό που χρησιμοποιείται, που μάλλον χρησιμοποιείται, λέει η πρόταση της Κομισιόν ότι για τα προϊόντα που περιέχουν βιοκτώνα θα πρέπει να αναφέρεται ε, στην ετικέτα και αριθμό αδειοδότησης. Θεωρούμε ότι είναι πιο χρήσιμο να περιλαμβάνει το όνομα του βιοκτόνου ή το, η ενεργή ουσία παρά ε, το νούμερο της αδειοδότησης. Αυτή η πληροφορία δεν είναι απαραίτητη για τον καταναλωτή, είναι απλώς ε, ε μια ε, επιβάρυνση για την επιχείρηση που την κατασκευάζει. Άρθρο 21, 17 και 18 και μάλλον 16, 17 και 18 θεσπίζονται τα επιστημονικά κριτήρια για την αξιολόγηση ενός βιοκτώνου. Στο 21 εντωμεταξύ ε, εισάγεται μία αξιολόγηση συγκεκριτικού τύπου. Αυτή την επιπρόσθετη αξιολόγηση για όλες αυτές που ήδη κανονικά προβλέπονται δεν γίνεται αναφορά στο άρθρο όταν και πότε θα πρέπει να την κάνει την αξιολόγηση αυτή η εταιρεία. Πρώτα έχουμε την αξιολο... πριν από την αξιολόγηση του 16, 17, 18 ή μετά. Αν αυτή η αξιολόγηση θα διατηρηθεί, θα πρέπει να μας πούνε και πότε πρέπει να την κάνει η επιχείρηση. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ κλείνουμε την εξέταση του 11 και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 12 της ημερησίας διάταξης. Για το σημείο 11, ο συνάδελφο Καρύμα ανέφερε τις προθεσμίε, δεν χρειάζεται να σε επαναλάβω. Λοιπόν, το 12 λέω, παρουσίαση μελέτη σχετικά με τα δίκτυα επόμενη γενιά. Έχουμε καλέσει δύο επισκέπτε που δεν ήρθαν ακόμα, ήρθαν. Για ένα λεπτό. nochmal. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, καθίσουμε όλε τι θέσει μα. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι βουλευτέ, έτσι. Ε, ναι. ε μεμονωμένοι.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 Thank you. It cannot be the beginning. It's the end normally. Ich meine, sonst unterhalten wir uns über was anderes Schönes. Αλλιώς να συζητήσουμε για κάτι άλλο ωραίο και ενδιαφέρον. Υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα με την παρουσίαση. wir haben jetzt auch noch ein technisches Problem. Das ist ja das Schöne, liebe Έχουμε και τεχνικό πρόβλημα. Αυτό είναι το ωραίο με τις παρουσιάσεις αυτές, αγαπητοί ε, συνάδελφοι. Mm Στο παρελθόν δεν υπήρχαν οι οθόνε. Ε, τώρα τις έχουμε και βλέπουμε τι μας παρουσιάσουν, αλλά αν δεν λειτουργεί όμως η τεχνολογία, χαθήκαμε. Και δεν είναι πρώτη φορά σήμερα που έχουμε προβλήματα. Es fällt mir ein. Wunderbar. Herr Scott Marcus weiß aber genau, was er gemacht hat. Ο κύριο Σκοτ Μάρκος ξέρει τι έκανε. Μπορεί να μας το πει και χωρί την παρουσίαση αυτή. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας χαιρετίζω εγκαρδιότατα. Κύριε Σκοτ Μάρκος και τον κύριο Τίτερ Χέλιξμαν, τους καλωσορίζω και τους δύο. Ξέχασα να σας το πω αυτό στη διασύνη μου. Θα χαιρόμαστε να μας παρουσιάζετε τις εργασίες σας. Έχουμε και γραπτά στοιχεία εδώ. Και αν μεταξύ η τεχνολογία κινηθεί, είμαι πεπισμένος ότι θα γίνει, θα δούμε και την παρουσία στις οθόνες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Äh, Ευχαριστώ, ξέρετε, κύριε Πρόεδρε. Αμερικανό είμαι, αλλά το λέω και στα γερμανικά. χαιρετίζω ιδιαίτερα την ιδιαιτότητα να είμαι παρόν εδώ σήμερα. Αυτό που θέλω να σας παρουσιάσω είναι η εξέλιξη των δικτύων στα δίκτυα της επόμενης γενιάς. Μια τάση που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μια τάση σύμφωνα με την οποία παραδοσιακά δίκτυα τηλεφωνίας να εξελίσσονται σε δίκτυα νέας γενιάς βασιζόμενες στις ίδιες ε, περίπου τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο. Το Internet Protocol IP λέμε. Υπάρχουν εξέλιξεις αυτές και ανάλογα με την εξέλιξη στην αγορά και όσον αφορά τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων και των διακανονιστών. Oh, there is. Thank you. Uh, I think thank you. Uh-huh. Well, uh, okay. I, I think we'll have a presentation in a minute. Ε, ε θα έχουμε την παρουσίαση εδώ, αλλά εντάξει, ε, μιλάω, δεν με νοιάζει. Μέσα πλαίσια αυτές θα δείτε κάποια παρουσίαση και υπάρχει μια συνολική παρουσίαση εξελίξεων σε 10 ευρωπαϊκές χώρες και σε όλο τον κόσμο λίγο. Ε, αυτό που είναι πάρα σημαντικό είναι ότι όταν περνάμε στα δίκτυα της νέας γενιάς βλέπουμε ότι οι παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ των υπηρεσιών και των άλλων δικτυών μεταφοράς έχει αποτύχει. Oh, it's, it's, up, it's okay up there. Oh, Okay, so I can just use space to form? Sorry. Okay, good. I think we actually have a presentation then. Έχουμε την παρουσίαση τώρα. Πολύ ωραία. Θαυμάσια. Για να δούμε. Αυτό που έχετε στην στην, ε, στην οθόνη σας δεν είναι παρά μόνο αυτό που έχω μπροστά μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές. Οι αλλαγές είναι ότι το ενιαίο δίκτυο έχει την δυνατότητα να προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες και προσφέρονται οι υπηρεσίες που δεν σχετίζονται και ε, σε δίκτυο. Παραδείγματο χάρη είναι ε, ηλεκτρονικές υπηρεσίες voice-over που δεν σχετίζονται με το δίκτυο. Εδώ έχουμε μία ένδειξη λοιπόν πώς ε, πραγματοποιείται ο ανταγωνισμός μέσα στα πλαίσια και μεταξύ δικτύων και ο ανταγωνισμός είναι ένας κύριος ε, ε, κινητήρας για τις αλλαγές. Μέσα στα πλαίσια των δικτύων υπάρχουν δύο βασικοί τόποι όπου λαμβάνει η χώρα μια σημαντική εξέλιξη. Καταρχήν στο πυρήνα των δικτύων και κατά δεύτερον στις, στα άκρα, στο σημείο επαφής. Σε πολλές περιπτώσεις εδώ έχουμε το voiceover και ε, αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές στο πυρήνα έχουν σαν στόχο να μειωθεί το κόστος και να επιταχυνθεί η προσφορά των υπηρεσιών. στο, στα άκρα το θέμα είναι η αλλαγή στις, σε τεχνολογία ινών. Ε, η επανάσταση που έχουμε βεβαίω είναι και οι προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστικέ αρχές. Ποιε είναι λοιπόν οι προκλήσεις από αυτέ τι ε, εξελίξει Είναι αρκετέ. Η πρώτη ήταν αυτή την οποία μόλι ανέφερα, οι αλλαγέ στην φύση του ανταγωνισμού εντός ενός δικτύου. Δεύτερον, η αλλαγή στην φύση του τι μπορεί να γίνει για το λεγόμενο τελευταίο χιλιόμετρο μέχρι τον λιανικό καταναλωτή. Ένα τρίτο ευρύτερο ερώτημα είναι το πώς θα υπάρξει ανάπτυξη του δικτύου. Ξέρουμε το πρόβλημα με την ε, παραδοσιακή ας πούμε ευρυζωνικότητα και βεβαίως υπάρχουν ε, ανάλογα ζητήματα όταν μιλάμε για οπτικές σύνες. Ένα τέταρτο μια τέταρτη σειρά ζητημάτων αφορά την μετάβαση στις διασυνδέσεις. Ιστορικά, τα δίκτυα τα οποία βασίζονταν σε κυκλώματα είχαν τεχνικές που βασίζονταν σε κυκλώματα με ένα σύστημα σημάτων 7 το λεγόμενο. Οπότε τώρα περνάμε σε ένα σύστημα IP κάτι το οποίο είναι, ε, σημαίνει ότι λογικό είναι να αλλάξουν και οι διασυνδέσεις. Ε, ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω εγώ καμία περίσταση στην οποία η εδρεωμένη εταιρεία σταθερής κινητής ε, έχει περάσει διασυνδέσεις ε, IP για το ενσωματωμένη την παραδοσιακή υπηρεσία φωνής για να το, προσφέρει αυτό στου ανταγωνιστέ. Αυτό δεν συμβαίνει και οι λόγοι σχετίζονται μάλλον με επιχειρηματικού και όχι τεχνολογικούς παράγοντες. Μία άλλη πρόκληση είναι κάτι το, για το οποίο έχετε ακούσει πολλές φορές σε σχέση με την ουδετερότητα του δικτύου. Δηλαδή έχουμε ανησυχίες για το ότι καθετοποιημένες επιχειρήσεις θα ευνοήσουν το δικό τους ε, το προϊόν, είτε αφορά περιεχόμενο είτε αφορά εφαρμογές, έναντι ε, των ανταγωνιστών. Θα το βρούμε, εν πάση περιπτώσει, στην παρουσίαση, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, η ουδετερότητα του δικτύου έχει πολλές διαφορετικές πτυχές, αλλά μία που συχνά αναφέρεται από τη μετάβαση στο IP είναι η ποιότητα της υπηρεσίας εντός του δικτύου. Σε ένα παραδοσιακό τηλεφωνικό δίκτυο είτε έχουμε σύνδεση είτε δεν έχουμε. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Σε ένα δίκτυο που βασίζεται στο πρωτόκολλο του ίντερνετ μπορούμε να έχουμε δίκτυα που είναι τόσο χάλια ώστε κατ' ουσίαν δεν έχουμε σύνδεση, αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα. Δηλαδή δεν είναι είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί η σύνδεση, υπάρχει, υπάρχουν και πολλές γκρίζες ζώνες μετάπτωσης της ε, ποιότητας. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες ίσως είναι επικερδές ε, για έναν ε, πάροχο του δικτύου που είναι καθετοποιημένος όσον αφορά τις υπηρεσίες του να ασκήσει τέτοιο έλεγχο. Είναι μεγάλη αυτή η συζήτηση στι Ηνωμένες Πολιτείες, λιγότερο τόσο στην Ευρώπη, αλλά είναι ένα ζήτημα που πρέπει να σκεφτούμε. Η μετάβαση επίσης στα δίκτυα νέας γενιάς ε, έχει δημιουργήσει και το ζήτημα της μεταβατικής περίοδου, καθώς ε, είναι πιο επίπεδα αυτά τα δίκτυα. Έχουν λιγότερη ιεραρχία, είναι, μοιάζουν λιγότερο με μια οργανωτική πυραμίδα. Ε, υπάρχουν λιγότερα αλλά και διαφορετικά σημεία με τα οποία συνδέεται κανείς στο δίκτυο. Αυτό είναι σημαντικό σε χώρες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια μετάβαση όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία. Υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα που πρέπει να αναφερθούν και σχετίζονται οπωσδήποτε πρότυπα και διαλειτουργικότητα. Πρέπει να συνεργάζονται όλες αυτές οι δυνατότητες. Διαχείριση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος ε, παίζει σημαντικό ρόλο εδώ πέρα για να έχουμε για να έχει ο κόσμος ε, συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και τέλος θα δείτε πώς πρέπει ε, να γίνεται αυτή η συζήτηση για, την, για το λειτουργικό διαχωρισμό και βέβαια όσοι έχετε ασχοληθεί με το σχετικό ε, νομοθετικό πακέτο αναθεώρησα, το γνωρίζετε. Δεν αφορά συγκεκριμένα τα δίκτυα νέα γενιάς, αλλά έχει τεθεί εκεί όπου γίνεται αυτή η μετάβαση στα δίκτυα νέα γενιάς, οπότε ίσως υπάρχει μια σύνδεση για να επανέλθουμε στα ζητήματα αυτά με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Αλλαγές στη φύση του ανταγωνισμού και πάλι το πλαίσιο το λειτουργικό αλλάζει, το ρυθμιστικό με συγχωρείτε αλλάζει με βάση το ποιο έχει ε, σημαντική δύναμη στην αγορά. Ελπίζουμε λοιπόν πως θα έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες ανταγωνισμού και σύν χρόνο να μειωθεί η ανάγκη ρυθμιστικής παρέμβασης. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και κάποιες στενοποί που δεν φαίνεται πως θα εξαφανιστούν σύντομα. Π.χ. αυτό το τελευταίο χιλιόμετρο στο σταθερό δίκτυο δεν θα εξαφανιστεί ε, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον. Επίσης ε, πράγματα του μονοπωλίου τερματισμού κλίσεων που συχνά οφείλεται στο ότι υπάρχει ένα μονοπόλιο και μόνο αυτό μπορεί να κάνει την κλίση προς ένα συγκεκριμένο νούμερο. Φαίνεται πως δεν θα εξαφανιστεί αυτό και ίσως να εμφανιστούν και νέες στενοποί. Οπότε, για τις ρυθμιστικές αρχές μακροπρόθεσμα ίσως υπάρχει μια ελπίδα για την μετάβαση, αλλά βραχυπρόθεσμα θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν και αυτοί και οι ε, πολιτικοί. Μία διαφάνεια θα ήθελα να φανεί. Δεν ξέρω. Α, ας ελπίσουμε. Στο α, ε, ρυθμιστικό πλαίσιο υπάρχουν ε, διαφορετικά πράγματα που μπορεί να γίνουν για την πρόσβαση στο τελευταίο ε, χιλιόμετρο, όπως λέγεται, από απλή μεταπόληση μέχρι bitstream, μέχρι αποδέσμευση τοπικού βρόχου, η μετάβαση στα δίκτυα νέας γενιάς λύνει κάποια προβλήματα, ειδικά όταν μιλάμε για οπτικές σύνες στην γειτονιά ή στο σπίτι. Ε, ακόμα και η δομημένη καλωδίωση γίνεται πάρα πολύ σημαντική. Μιλάμε για στενοπούς τα τελευταία 100 μέτρα Επίσης ε, λύσεις που έχουμε όπως VDSL ή ίνες στον κόμβο σημαίνει πως πηγαίνει η Ines στον ε, πελάτη από πλευράς διανομής. Οπότε ε, αυτό σημαίνει πως εξυπηρετούνται λιγότεροι πελάτες και υπάρχουν σοβαρές αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο. Έχουμε κάνει μελέτες για την οικονομία Ανάπτυξη αυτών των δικτύων και έχουμε άρα κάποιες ανησυχίε για την ευρεία ανάπτυξή τους. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι το κόστος το οποίο σημαίνει είναι τέτοιο ώστε δεν θα έχουμε κάλυψη όλης επικράτειας οποιοδήποτε κράτης μέλους μόνο με βάση δυνάμεις αγοράς. Ε, όταν μιλάμε για οπτικές ίνες. Δεύτερον, ε, εντός ενός κράτους μέλους αυτή τη στιγμή ξεκινήσει κάποιος, δεν ανάγκη η κυρίαρχη εταιρεία, ε, είναι απίθανο μια δεύτερη εταιρεία μετά να καλύψει ολόκληρη την επικράτεια. Δεν έχει επιχειρηματική λογική. Αυτές είναι οι συνέπειες. Η έκθεση καλύπτει κάποιες, ε, προοπτι... κάποιες ε, πρωτοβουλίες που υπάρχουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη βέβαια είναι το πακέτο αυτό της αναθεώρησης νομοθεσίας και υπάρχουν αρκετά πράγματα που ε, έχουν σχέση εδώ πέρα, π.χ. το να αναγνωρίσουμε ότι οι εταιρείε οι οποίες αναπτύσσουν αυτά τα δίκτυα αναλαμβάνουν υψηλότερο κίνδυνο και πρέπει αυτό να αντικατοπτρίζεται και στο κέρδος το οποίο τους επιτρέπεται από την επένδυσή τους υπάρχει η παρατήρηση πως ε, οι υποδομές αυτές ε, και οι καλωδιώσεις των κτηρίων πρέπει να ληφθούν υπόψη για πρώτη φορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι καινοτομίες. Όπως σημειώσαμε στο παρελθόν υπάρχει μια γενική ενδυνάμωση και δυνατότητα των κρατών μελών για να εφαρμόσουν τον λειτουργικό διαχωρισμό, αλλά μόνο σε ακραίε περιπτώσεις, που κατά την άποψή μας πάλι είναι λογικό. Ένα άλλο θέμα είναι οι κατευθυντήριες ε, γραμμές κομισιών για τις κρατικές ενισχύσει που διακρίνουν μεταξύ μαύρων, γκρίζων και άσπρων περιοχών, δηλαδή αυτές όπου θα έχουν πλήρη κάλυψη, ελάχιστη κάλυψη και αυτές που καλύπτονται μόνο από έναν πάροχο από μία κάλυψη αυτές τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες και υπάρχει το ζήτημα του ποια θα είναι η κατάλληλη κρατική ε, παρέμβαση όταν έχουμε μόνο ένα δίκτυο. Τέλος, βλέπουμε για, την, για τον δροματισμό κλήσεων σταθερών και κινητών που έχει ένα ρόλο στον χώρο αυτών στο παρελθόν είχαμε εργαστεί για την Κομισιόν και είχαμε προτείνει να μειωθεί το τέλος τερματισμού κλήσεων γιατί θα έφευγε έτσι ένα εμπόδιο για την μετάβαση στις διασυνδέσεις ε, για να μεταβούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο θα βασίζεται σε IP και φαίνεται πως η σύσταση αυτή ανεξαρτήτως του ε, μηχανισμού ε, φαίνεται πως οδηγεί τα τέλη τερματισμού σε ένα λογικό ύψο. Οπότε φαίνεται ότι κολλάει και συζήτηση για τα δίκτυα νέα γενιά. Έχουμε κάνει και κάποιε άλλε συστάσει στην εκθεσή μα και ελπίζω να τη διαβάσετε λεπτομερώ. Το πρώτο αφορά το πακέτο αναθεώρηση που εκκρεμεί. Θεωρούμε γενικά πω η στάση για τα δίκτυα νέα γενιά ε, δεν ε, ήταν οι κατάλληλε. οπότε η πρώτη σύσταση που κάναμε ήταν ε, περάσει αυτό το πακέτο και φαίνεται πως ε, έγινε δεκτή η πρώτη μας ε, σύσταση και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Η δεύτερη σύσταση είναι πως ίσως ήταν καλό να γίνει καλύτερη χρήση των λεγόμενων υποεθνικών αγορών. Το ρυθμιστικό πλαίσιο πάντα επέτρεπε τον ορισμό της αγοράς στο πιο κατάλληλο επίπεδο, αλλά αναγνωρίζεται πλέον πως η χρήση αγορών που καρύπτουν όλη την επικράτεια του κράτους μέλους δεν είναι ο μόνος τρόπος που είναι δυνατός. Λίγα κράτη-μέλη έχουν μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση και είναι πιθανόν η πρόσβαση στην... στα δίκτυα νέας γενιάς ε, να οδηγήσει σε πιο διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά εντός της επικράτειας και άρα να δημιουργηθούν διαφορές ή μάλλον να οδηγηθούμε σε υποεθνικές αγορές. Τρίτη σύσταση είναι να πάρουμε την ε, σύσταση της Κομισιόν για την πρόσβαση στην ε, νέα γενιά, στα δίκτυα νέας γενιάς, να γίνει όσο το δυνατόν πιο πλήρης αυτή και φαίνεται πως ε, πράγματι Εντάξει, είναι σε γενικέ γραμμέ καλή. σω εκεί που μιλάμε για πολλαπλέ είναι, είναι κάποιο διαφορετικά τα πράγματα όπω νομίζαμε, αλλά γενικά πηγαίνει σωστή κατεύθυνση και πρέπει να ολοκληρωθεί. Πάρα πολλέ από τι συστάσει μα ε, αφορούσαν το πώ ε, θα έχουμε πρόσβαση και ευρυζωνικότητα γενικά στα νέα δίκτυα σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Ποιε είναι οι σωστέ πρωτοβουλίες. Τι συστάσεις αυτέ, η πρώτη μας ήταν μια καλύτερη αντίληψη του κόστους και του ωφέλους της πρόσβασης ε, νέας γενιάς. Αρκετές μελέτες αξιολόγησαν το κόστος και το όφελος της ευρυζωνικότητας, αλλά ελάχιστα λίγα ποσοτικά δεδομένα είχαμε για το πραγματικό κόστος και όφελος, ειδικά μακροοικονομικά ε, όσον αφορά ε, μακρονομικά ειδωμένα για την ε, πάρα πολύ μεγάλη αύξηση της ε, ταχύτητας πρόσβαση. Και νομίζω πως, όπως είδαμε και εγώ και ο συνάδελφος ο κύριος Τίτερ εδώ πέρα, η γενική άποψη είναι πως φαίνεται καλό πράγμα, αλλά δεν υπάρχει μια ποσοτικοποίηση και χρειάζεται μια πιο σοβαρή μελέτη. Και αν υποθέσουμε πως τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα θα είναι θετικά όπως αναμένουμε, νομίζω πως καλό θα είναι να κοιτάξουμε καλύτερα τις ε, πρωτοβουλίες ε, του δημόσιου τομέα για να προωθηθεί η πρόσβαση νέας γενιάς και το δε πακέτο αναθεώρηση που κοντεύει να ολοκληρωθεί ασχολείται με την ρυθμιστική πτυχή της ε, πολιτικής του δημοσίου, αλλά υπάρχουν και άλλες πτυχές αυτής της πολιτικής και ειδικά εάν γίνει μια αξιολόγηση εξ άντε όσον αφορά τον αντίκτυπο, να δούμε ποιο είναι πάλι το κόστος όφελος, το τι, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν και έχοντας αυτά τα μέσα νομίζουμε πως ε, υπάρχει μια συζήτηση που πρέπει να γίνει πολιτική στην Ευρώπη για το ποιοι είναι οι στόχοι κάτι σαν το 2010 e ή κάτι σαν την ατζέντα ε, της Λισαβόνας. Ποιος είναι ο στόχος, ε, τι πρέπει να καλύψουμε με τα, νέα, τα δίκτυα νέας γενιάς, με ποια ταχύτητα, σε ποιο χρονοδιάγραμμα. Δεν φτάνει το πακέτο το αναθεωρητικό εκεί. Κάποιες χώρες έχουν τοποθετηθεί και η Ευρώπη δεν ε, παίζει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη τέτοια πρόσβασης δικτύων νέας γενιάς. Η Ευρώπη πήγε πάρα πολύ καλά γενικά όσον αφορά την ευρυζωνικότητα, αλλά αν δούμε τις οπτικές σύνες υπάρχουν ε, η Ιαπωνία, η Κορέα, η ΙΠΑ και άλλα μέρη όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Σιγκαπούρη που μπορούν να φτάσουν και αυτά σε ένα τέτοιο επίπεδο. Τώρα, ε, ακριβώς θεωρούν πως χρειάζεται μία ανάλυση του κόστου και του ωφέλου, γιατί δεν είναι σαφές το εάν είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει την Ευρώπη ή όχι. Θεωρούμε λοιπόν πως ε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν τα ποσοτικά δεδομένα για να το κρίνουμε. Υπάρχουν και κάποιες άλλε συστάσεις εντό τη Θεωρούμε πως πρέπει να γίνει μια πιο σοβαρή ε, αξιολόγηση της ε, τακτικής ε, τιμολόγησης και διατήρησης. Ε, κάτι το οποίο ζήτησαν πολλές, πολλά θεσμικά όργανα, μεταξύ των οποίων και η Ένωση των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών. Εγώ βέβαια είμαι Αμερικάνος γνωρίζω πολύ καλά αυτή την τακτική, θεωρούν πως είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Το να πάμε επίσης προς μια διασύνδεση IP δεν πως είναι κάτι που απαιτεί κάποια ιδιαίτερη πρωτοβουλία, αλλά είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για το αν προχωράει όπως θα ήθελαν. Είναι πολύ ε, αργότερη ταχύτητα από αυτή που αναμένονταν ακόμη και πριν από 10 χρόνια. Και τέλος, όσον αφορά το φάσμα, πρέπει να συνεχίσουμε να αναζητούμε ευκαιρίες για διάθεση φάσματος ε, υψηλής ποιότητας για σταθερή ή κινητή ευρυζωνικότητα. Γιατί μας φαίνεται λογικό πως ε, δεν θα καλύψει 100% της επικράτειας των κρατών μελών ε, οι οπτικές σύνες, οπότε θα πρέπει κάπου αλλού να είναι ασύρματη η λύση και όπου μπορεί να απελευθερωθεί φάσμα αξίζει να το εξετάσουμε σοβαρά. Δεν προτείνουμε εδώ πέρα μια αλλαγή πολιτικής. Νομίζουμε πως αυτό κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Απλά προτείνουμε να περάσουν γενικά στην, στην επόμενη γενιά και με το να γίνει αυτό θα γίνει ακόμη πιο σημαντική αυτή η κίνηση. Αυτά και τελείωσα. Ε, είμαι σίγουρος ότι θα έχετε ερωτήσεις. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρκος, πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας, <coughs> ακόμα και χωρίς παρουσίαση στην οθόνη. Υπάρχουν ερωτήσεις? Εάν όχι, να δώσουμε το λόγο στην κομισιον Κύριος, ε, κύριε Ρότφορ, θέλετε δύο-τρεις προτάσεις να πείτε για το θέμα και αν κάποιοι συνάδελφοι έχουν ερωτήσεις να τις ακούσουμε, αλλιώς θα συνεχίσουμε. Thank you very much, Ευχαριστώ Πρόεδρε και σα ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να σχολιάσω πολύ σύντομα. Θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή Ιντρα που ανέθεσε την μελέτη αυτή. Πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή μελέτη. Δείχνει μια σωστή εικόνα, νομίζουμε, τη κατάσταση σε σχέση με τα δίκτυα νέας γενιάς. Ε, έχουμε προβλήματα με κάποιε λεπτομέρειε, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνουμε εδώ. Είναι φυσιολογικό κάτι τέτοιο. Πρέπει να σα αναρωτιέμαι. Το Void είναι μια υπηρεσία που μπορεί να προσφερθεί εδώ. Ε, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η μελέτη αυτή εξετάζει τις συστάσεις της Κομισιόν σαν θετικές και χαιρετίζουμε το δήλωση ότι η σύσταση αυτή όταν υποβληθεί θα δώσει επαρκή σαφήνια ε, σαφήνεια για πολλές ε, οργανώσεις το τονίζουμε αυτό, συμφωνούμε. Αυτό το θέμα εξετάζεται και μέσα στα πλαίσια των καθημερινών γραμμών για ε, τις κρατικές βοήθειες. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες διστάσεις εδώ, αναγνωρίζουμε πολλές από αυτές. Ε, θέλουμε βέβαια να υιοθετηθεί η δέσμη αναθεώρηση των γρηγορότερων δυνατών. Λαμβάνουμε υπόψη μας τις συστάσεις στα υποεθνικά ε, δίκαια, στις υποεθνικές αγορές, αυτό είναι κάτι που συμπεριλαμβάνεται στην αναθεωρημένη εκδοχή της σύστασης μετά από την δεύτερη δημόσια διαβούλευση. Πιστεύουμε ότι μέσα στα πλαίσια του I2010 θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό που είχατε προτείνει και εσείς σχετικά η μεγαλύτερη παρουσίαση, ακούσαμε τις ε, παρατηρήσεις που είχαν γίνει εδώ στο Κοινοβούλιο για τη δέσμη ε, των μέτρων για τις ε, καθολικές υπηρεσίες και θα δούμε πώς μπορούν αυτές να χρησιμοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθεί η ευρυζώνη για όλους. Αυτό είναι τα κύρια συμπεράσματα που, στο οποίο καταλήγω έχοντας ακούσει την παρουσίαση και σας ευχαριστώ για μια φορά που αναθέσατε την μελέτη αυτή. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο που να ζητάει το λόγο. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε το σημείο αυτό τη ημέρα τη διάταξη. Σα ευχαριστώ κύριε Μάρκο. Ήταν όλα φαίνεται πολύ σαφή και ακριβή και γι' αυτό δεν χρειαζόταν συμπληρωματικέ ερωτήσει. Σα ευχαριστώ πολύ που ανεματοποίησατε και το τεχνολογικό πρόβλημα χωρί ε, πρόβλημα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου. Περνώ στο σημείο 13 και 14 τη ημέρα τη διάταξη. Η επόμενη συνεδρίαση προβλέπεται 2 και 3 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρουμε αν θα λάβει χώρα όμως. Γιατί ίσως εκείνη την εβδομάδα θα λάβει ακριβώς ε, χώρα η ακρόαση των επιτρόπων. Αλλά δεν ξέρουμε ποτέ αν τα σχέδια θα πραγματοποιηθούν. Θα σας ε, πρότεινα λοιπόν να προβλέψετε τις δύο αυτές ε, ημερομηνίες. Ελίσως την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου έχουμε τέσσερις συνεδριάσεις για να ακούσουμε τους επιτρόπους. Τώρα κατά πόσο αυτό θα γίνει αυτές τις δύο μέρες, άλλες μέρες δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά όλα θα αποφασιστούν τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που άντεξαν μέχρι τώρα. Ε, πολύ επίπονοι συναδελφοί άντεξαν εδώ όλα την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ και πραγματικά να τελειώσουμε λίγο νωρίτερα ήταν καλό για όλους.